Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να αρχίσουμε. good morning. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Παρατηρήσεις, Εγκρίνεται λοιπόν. Ανακοινώσεις. Η πρώτη μου ανακοίνωση έχει να κάνει με την ακύρωση συνεδριάσεων εξαιτία των ακροάσεων που θα έχουμε με τους υποψήφιους επιτρόπους. Οπότε, οι συνεδριάσεις μας 13 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου ε, συγγνώμη, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου ε, αναβάλλονται προκειμένου να μπορέσουμε να οργανώσουμε τις ε, ακροάσεις αυτές. Τώρα ποιο θα είναι ο ρόλο τη ΕΝΒΗ, πώ θα οργανωθούν αυτές οι ακροασει. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν, για την Επίτροπο Υγείας, και επίσης θα οργανώσουμε από κοινού με την Επιτροπή Αλίας την ε, ακρόαση για την Επίτροπο την Αρμόδια για την Αλία και τους ωκεανούς. Και είμαστε και προσκεκλημένοι επίσης σε άλλες ακροάσεις στην γεωργία, τις μεταφορές, την ενέργεια, την προστασία των πολιτών και στον κύριο Ντομπρόφσκι που είναι οικονομία για τους ανθρώπους, κάπως έτσι δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο. Οπότε έχουμε διάφορες ακροάσεις στις οποίες θα πάμε. Είτε ως επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή, είτε ως συνδεδεμένη, είτε ως προσκεκλημένη. Και θα πρέπει να θέσουμε διάφορες ερωτήσεις. Θα πρέπει να οργανωθούμε και αυτό θα αποφασιστεί σήμερα το πρωί στη συνεδρίαση των συντονιστών που έχουμε σήμερα στο τέλος του πρωινού. Και εννοείται θα σας ενημερώσουμε για το πώς θα οργανωθούμε τελικά. Η τελευταία μου ανακοίνωση έχει να κάνει με αλλαγές στη γραμματεία. Γιατί η Σαντελιέτε Κάρετ έφυγε από την γραμματεία, πήγε στον πρόεδρο Σασόλιο που θα είναι η υπεύθυνη για τον οριζόντιο συντονισμό εκεί. Συγχαρητήρια λοιπόν. Είναι ωραία, βέβαια να έχουμε έτσι κάποιον από την ε, η γραμματεία της ΕΝΒΗ. Επίσης μην ξεχάσετε στις 2.30 ότι θα ψηφίσουμε. Γι' αυτό να έχετε τις κάρτες σας μαζί. Αυτά για τις ανακοινώσεις όσον αφορά τις εστάσεις των συντονιστών από την προηγούμενη συνεδρίαση κυκλοφόρησαν ηλεκτρονικά. Οπότε αν δεν έχετε κάποια συγκεκριμένη παρατήρηση μπορούμε να προχωρήσουμε. Και περνάμε στην αυτή καθεαυτή μερίσια διάταξη και όπως γνωρίζετε θα έχουμε πρώτα απ' όλα μια αλλαγή. Τα σημεία 4 και 5 θα αλλάξουν σειρά. Πρώτα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά ΕΦΣΑ. Πρώτα το σημείο 5 δηλαδή και μετά το σημείο 4. Συνεπώς, θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Υγείας. Όσον αφορά τον κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού 546 του 2011, όσον αφορά την αξιολόγηση του αντικτύπου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μέλισσες. Ποιο είναι το πλαίσιο είναι ότι οι πολιτικές ομάδες ζήτησαν, κυρίως οι πράσινοι και η γκουε, να γίνει αυτή η συνάντηση και το αποφασίσαμε στους συντονιστές στις 4 ε, Σεπτεμβρίου όντως να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την ΕΦΣΑ μετά για να ξέρουμε ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πού βρισκόμαστε και να δούμε τελικά τι αποφάσεις θα πάρουμε. Οι συντονιστές λοιπόν αποφάσισαν για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων, διότι υπάρχει δυνατότητα οι ευρωβουλευτές και το ΕΛΚ είτε να δεχτούν είτε να απορρίψουν αυτή την πρόταση της τροποποίησης. Και η προθεσμία είναι 27 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή δηλαδή. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων σήμερα, πριν εκπνεύσει δηλαδή η προθεσμία, για να υποβάλουμε αντίρρηση εφόσον θέλουμε να μην προχωρήσει η τροποποίηση αυτή. Λοιπόν, είπαμε 27 είναι η προθεσμία. Και μετά αν υπάρχουν αντιρρήσεις θα πρέπει να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και εφόσον ε, ψηφιστεί η αντίρρηση αυτή θα πάμε στην Ολομέλεια. Και για την Ολομέλεια η προθεσμία είναι Οκτωβρίου. Στο Στρασβούργο δηλαδή, στην Ολομέλεια, θα συνεχίσουμε εάν ξεκινήσει αντίρρηση από πλευρά σας. Αυτά για να γνωρίζετε Πώ έχουν τα πράγματα και γιατί οι συντονιστέ αποφάσισαν να γίνει σήμερα αυτή η ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο στον Ταν Σέμπερενς που είναι υπεύθυνο του τμήματο ε, φυτοπροστασίας και παριστοκτόνων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και καλημέρα Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω ότι η προστασία των μελισσών και της επικονίασης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην γεωργία, αλλά και για τη φύση συγχρόνως. Επίσης υπενθυμίζω ότι οι δραστικές ουσίες και τα προϊόντα φυτοπροστασίας ετίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο εφόσον προηγουμένως έχει υπάρξει επιστημονική ε, έγκριση ότι είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον, ακόμα και όσον αφορά τις επιπτώσεις δηλαδή που έχουν και στα έντομα. Για να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι αυτές οι επιστημονικές αξιολογήσεις γίνονται αρμονισμένα στις χώρες μέλη και στην ΕΦΣΑ, υπάρχουν κάποια έγγραφα όπως η κατευθυντήρια γραμμή για την αξιολόγηση που έχουμε για τις μέλισσες που είναι από το 2002, όπως επίσης και ένα άλλο αντίστοιχο του 2013 της ΕΦΣΑ μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έγγραφο κατευθυντηρίων γραμμών ε, τίθεται σε εφαρμογή εφόσον το έχουν ζητήσει οι χώρες και η Επιτροπή για τα τρόφιμα και για τις ζωοτροφές. Και μόνο τότε πρέπει να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης δραστικών ουσιών ή για την ανανέωση τέτοιων εγκρίσεων. Τώρα, δυστυχώς, ακόμα και μετά από πέντε χρόνια συζητήσεων ε, για το συγκεκριμένο έγγραφο προς Ανατολισμού, μόνο λίγες χώρες συμφώνησαν να θέσουν σε εφαρμογή άλλε Εν μέρη το έθεσαν σε εφαρμογή και πολλοί έχουν ζητήσει πλήρη αναθεώρηση πριν τεθεί σε εφαρμογή. Για να σταματήσει λοιπόν αυτό το αδιέξοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, πρότεινε από πέρυσι, ξεκίνησε να εφαρμοστούν πρώτα τα τμήματα των κατευθύνων γραμμών του 2013 που έχουν να κάνουν με τους οξύ κινδύνους για τις μέλισσες, επειδή υπήρξε στήριξη επ' αυτού από τις χώρες μέλη και να ζητήσουμε από την ΕΦΣΑ να αναθεωρήσει τα άλλα σημεία που έχουν να κάνουν με τα χρόνια προβλήματα, που έχουν να κάνουν επίσης και με τις ε, μεμονωμένες ε, μέλισσες που δεν ζουν σε απικίες. Η αναθεώρηση αυτή θα λάβει χώρα κυρίως νέα ε, επιστημονικά δεδομένα, ε, τα οποία έχουμε μετά το 2013. Και υπάρχουν πολλά από αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση ζήτησε από την ΕΦΣΑ να διασφαλίσει ότι αυτή η διαδικασία αναθεώρηση θα λάβει υπόψη τη όλου του ενδιαφερόμενου, ώστε ε, τα νέα δεδομένα να γίνουν αποδεκτά από όλου, τέλο πάντων από τη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών μελών. Η ΕΦΣΑ θα εξηγήσει στη συνέχεια πώς θα προχωρήσει η διαδικασία αυτή, αλλά ήδη από τώρα μπορώ να σας πω ότι η πρώτη συνάντηση που είχαμε με τις ενδιαφερόμενες πλευρές της χώρες μέλη θα λάβει χώρα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Το σχέδιο κανονισμού που συζητάμε σήμερα έχει ως ε, στόχο να τροποποιήσει τις ε, ομοιόμορφες ε, διατάξεις και πρόκειται κυρίως για τα στοιχεία εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν με τους οξύς κινδύνους για τις μέλισσες. Εφόσον εγκριθεί, οι αλλαγές των κριτηρίων θα βοηθήσουν στην εφαρμογή των σημείων του γράφου του 2013 της ΕΦΣΑ για να λυθούν υπόψη και άλλοι οδοί που βρουν αρνητικά για τις μέλισσες, όπως είναι ψεκασμοί με σπρέι και άλλοι. Και έχει καταλήξει αυτά η ΕΦΣΑ μέσα από επιτόπιες μελέτες ή εν μέρει επιτόπιες μελέτες. Όσον αφορά λοιπόν την οξία τοξικότητα, σας είπα τώρα για τις χρόνιες περιπτώσεις. Θα συνεχίσουν τα πράγματα όσοι έχουν μέχρι τώρα. Ο κανονισμός ο οποίος λέει τι δεδομένα χρειάζονται, ήδη σήμερα απαιτεί δοκιμές για την χρόνια τοξικότητα στην οποία μπορεί να εκτεθούν οι μέλισσες. Και τα δεδομένα που έχουμε υπάρχουν στους φακέλους εφαρμογής και λαμβάνονται υπόψη από την ΕΦΣΑ. Στα συμπεράσματα στην διαδικασία peer review η ΕΦΣΑ αξιολογεί τα δεδομένα βάσει των σημερινών κατευθυντηρίων γραμμών του 2002 δηλαδή, αλλά συμπεριλαμβάνει και μια ανάλυση βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών του 2013. Οι πληροφορίες αυτές είναι στη διάθεση των χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να η υπόψη στη μόνιμη επιτροπή. Τώρα για την έγκριση της ε, μιας δραστικής ή Παράταση της έγκρισης πρέπει να σεβόμαστε την νομοθεσία και οι αποφάσεις ε, δηλαδή ε, προς το παρόν να λαμβάνονται βάσει των κατευθύνων γραμμών του 2002, αλλά βάσει της ανάλυση ε, της ΕΦΣΑ και βάσει των νέων στοιχείων που έχουμε για κενά ή νέα επιστημονικά στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα λάβει υπόψη της και ήδη έχει ξεκινήσει είτε με απαιτήσει για νέα δεδομένα, είτε με μια νέα διαδικασία βάσει του άρθρου 21 του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως κάναμε και κατά το παρελθόν για τα νεονικοτιδή το 2013. Στην πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε στην απόφασή του στην περίπτωση που έχει να κάνει με τους περιορισμούς που εγκρίθηκαν για τα τρία νοικοτινοειδή, ότι η έγκαιρη αναθεώρηση, οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να ε, ληφθούν υπόψη παρόλο που δεν έχουν εγκριθεί από τη μόνιμη επιτροπή. Συνεπώ, για να ολοκληρώσω, υπογραμμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λυπάται που οι χώρες μέλη δεν ήταν έτοιμες να στηρίξουν τα περισσότερα από τα όσα προτείναμε εμείς στον κανονισμό δεν ήταν δυνατόν να πετύχουμε πλειοψηφία για να στηριχτεί η εφαρμογή όλων των στοιχείων των κατευθυντήριων γραμμών του 2013 πριν γίνει αναθεώρηση. Η έγκριση του σχεδίου κανονισμού που βρίσκεται ενώπιόν σα είναι ένα βήμα προς τα μπρο και πρόκειται για μια βελτίωση όσον αφορά ε, τους οξύ κινδύνου για τις μέλησει, που είναι κάτι καλύτερο από το να μην γίνεται τίποτα όπως δεν γινόταν τίποτα τα τελευταία πέντε χρόνια. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι εφόσον ολοκληρωθεί η αναθεώρηση που ζητήσαμε από την ΕΦΣΑ και έχει ήδη ξεκινήσει, τα υπόλοιπα στοιχεία, δηλαδή μια καλύτερη μεθοδολογία ε, για την χρόνια τοξικότητα και τα όσα ξέρουμε για τις αγρομέλισσες τους βομβίνους δηλαδή ή για τις μέλισσες εκτός ε, απικιών μπορούν να προχωρήσουν προσβλέπουμε τώρα στην πλήρη εφαρμογή στη συνέχεια των νέων κατευθυντήριων γραμμών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα συζητήσουμε τον εξή τρόπο. Θα ξεκινήσουμε με τις δύο ομάδες. οι οποίες ζήτησαν και τη συζήτηση ε, και εν συνεχεία θα περάσουμε στο Catch the Eye. Εάν θέλετε το λόγο να μας πείτε. Θα ξεκινήσουμε με δύο λεφτά για τους πράσινους και δύο λεφτά για τον κύριο Μπιόν από την Γκουέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν που προσπάθησε να εξηγήσει τι συνέβη. Παραμένουν κάποια ερωτήματα ακόμα. Η ΕΦΣΑ είχε τις κατευθυντήριες γραμμές από το 2013 και οδήγησαν στην απαγόρευση αυτών των τριών νεονικοτινοειδών το 2013. Αυτό το επιβεβαίωσε και το δικαστήριο. Πέρυσι όμως, 16 κράτη-μέλη είχαν αντίρρηση σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμέ που αφορούσαν τις χρόνιες επιπτώσεις. Αυτό που προτείνεται τώρα είναι να ασχοληθούμε με τις οξύες επιπτώσεις και να καθυστερήσουμε την ε, αντιμετώπιση των χρονίων. Έτσι δημιουργείται διπλά πρότυπα. Γιατί τα τρία νεονικοτινοειδή τα αντιμετωπίσαμε τις κατευθυντρίες γραμμές το 2013, απαγορεύτηκαν και τώρα επιβεβαιώνεται ότι θα, θα εξετάζουμε μόνο τις οξύες περιπτώσεις. Και ελπίζεται ότι η αναθεώρηση θα γίνει έγκαιρα, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουν κάποτε και οι χρόνιες περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής ε, βλέπουμε καθυστέρηση πάνω στην καθυστέρηση. Αυτό το θέμα το έχουμε στην ατζέντα μας από το 2009. Γιατί πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα καταφέρουμε, πώ εξηγείτε ότι, εξηγούμε, ότι έχουμε τώρα διπλά πρότυπα, έχουμε τι κατευθυντήριες του 2013, απαγορεύτηκαν τα τρία νεονικοτινοειδή. Τώρα λέτε όμω ότι θα ασχοληθούμε μόνο με τι οξύε περιπτώσει, Ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τι χρόνιες περιπτώσει, γιατί το λέει η νομοθεσία ότι πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε και το πιο σημαντικό είναι γιατί η Κομισιόν δεν έφτασε σε πολιτικό επίπεδο όλα τα εξετάσατε σε επίπεδο ομάδα εργασία. Πώ θα ξέρουν οι άνθρωποι εδώ ότι η δική του χώρα, α πούμε, είχε αντίρρηση να αντιμετωπίσει τι χρόνε περιπτώσει. Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, πολλέ από αυτέ τι χώρε. Ενώ ξέρουμε ότι σε δημόσιο επίπεδο έχουν άλλη συζήτηση. Η Κομισιόν θα μπορούσε να είχε προτείνει τι κατευθυντήριε γραμμέ του 2013 και να είχαν συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο. Για να είμαι σίγουρο ότι καμία από αυτέ τι χώρε δημόσια θα μπορούσε να είχε πει εμεί δεν θέλουμε να το, μάλλον να, να βγει και να το πει αν ήθελε, αν μπορούσε, α, εμείς δεν θέλουμε να υπερασπιστούμε τις μελισσές μας, ας πούμε. Γιατί το γεγονός ότι δεν έβαλατε το θέμα αυτό ε, στο πολιτικό επίπεδο, αποδυναμώνει τα, τα πράγματα, δεν αντιμετωπίζει τις χρόνιες περιπτώσεις, γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει το Κοινοβούλιο να, να αναλάβει δράση τώρα. ε, κυρία Μπιόργκ, από τους Πράσινους. Ε, από την ΚΟΕ. Ε, το όνομά μου σημαίνει αρκούδα στα σουηδικά. Όπω είπε και ο προηγούμενο ομιλητή, αυτό το σημερινό τι σημαίνει. Ότι δεν κάνουμε ό,τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να σταματήσουμε την καταστροφή των μελισσών. Δείχνει ότι οι μεγάλες ε, εταιρείε ε, χημικών κατάφεραν να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία με συνεχείς καθυστερήσεις, αλλά εμείς θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν θα σταματήσουμε και ότι θα έχουμε καλύτερες στο μέλλον δοκιμές. Η χρόνια τοξικότητα και οι, υπο... και θανατηφόρες επιπτώσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Επιπλέον, ένα επιπλέον ερώτημα σε σχέση με τα περσινά. Πώς θα με εξασφαλίσει η Κομισιόν ότι οι δοκιμές που θα προκύψουν μετά από αυτή την αναθεώρηση δεν θα αποδυναμώσουν τα επίπεδα που προτείναμε το 2013. Που τα, πρότειναν, που τα πρότεινε η ΕΦΣΑ δηλαδή με τις δοκιμές τότε. Όπως υπόθηκε είναι πολιτικό το θέμα. Δεν νομίζω ότι αν ήξερε ο κόσμος τι παίζεται, ποιες χώρες είναι αντίθετες, ε, θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη πίεση να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα. Γιατί ο κόσμος ξέρει ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, η Άνια ήρθε, μόλις ήρθε. Έχουμε συνεργαστεί πάνω σε αυτό το θέμα. Θα ήθελε ίσως να προσθέσει κάτι. Πάμε στο Eye. Ένα λεπτό ο καθένας, παρακαλώ. Οι σοσιαλιστές. Κυρία Γκούδελον, ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ Κομισιόν. Συμφωνώ με τους δύο προλαλήσαντες. Δεν θέλουμε καθυστέρηση πάνω στην καθυστέρηση. Θέλουμε αντίθετα πολλαπλές δράσεις, τη μία μετά την άλλη. Οι πολίτες των κρατών μας το θέλουν επίσης. Ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση, ότι υποφέρουν οι μέλησεις από τα χημικά, από τα φυτοφάρμακα και πεθαίνουν. Είναι τεράστιο πρόβλημα την κοινωνία μας οι μέλισσες και οι επικονιαστές είναι σημαντικές για τα οικοσυστήματα. Δεν χρειάζεται να σας το πω, το ξέρετε. Γιατί η Κομισιόν λοιπόν δεν κάνει κάτι για να προστατεύσει τα ίδια αυτά. Επί δεκαετίες είδαμε ότι οι πληθυσμοί αυτοί σταθερά μειώνονται σε όλη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι τεράστιο θέμα. Θα επηρεάσει τη ζωή μας και το μέλλον μας. Αλλά δεν χρειάζεται να υποκύψουμε. Αν χρησιμοποιήσουμε την επιστήμη και τους κανόνες, μπορούμε να τις προστατεύσουμε τις μέλισσες και αυτό το ξέρουμε. Η απαγόρευση των νοικοτινοειδών είναι ένα παράδειγμα όπου χρησιμοποιήθηκε μια καλή επιστημονική διαδικασία με σωστό τρόπο. Και το ξέρουμε, που δεν κάνουμε κάτι άλλο. Είναι παράλογη η κατάσταση. Έχουμε το έγγραφο με τις ε, κατευθυντήριες γραμμές, αντί να το χρησιμοποιήσουμε όμως και να έχουμε μια πλήρη μεθοδολογία, το αγνοούμε. Και τώρα υποτίθεται η Κομισιόν κάνει μια αναθεώρηση του εγγράφου, που σημαίνει ότι μέχρι το 2021 αυτή η μεθοδολογία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρησιμοποιηθεί. Θέλω λοιπόν μια σαφή απάντηση από την Κομισιόν. Ε, το έγγραφο για, την, ε, για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ε, μέλισσες θα χρησιμοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η αναθεώρηση ή δεν θα, θα συνεχίσουμε έτσι, δεν θα προστατεύουμε τις μέλησες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ήσασταν οι μόνοι από τους σοσιαλιστές, ήσασταν λίγο παραπάνω χρόνο. Οι υπόλοιποι όμως, ειδικά οι πράσινοι και ε, τα μέλη της Renew, ένα λεπτό αυστηρά. Chris Davis, Renew. I want to know... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξέρω ποιο έχει την ευθύνη εδώ. Γιατί ε, το έγγραφο καθοδήγησης της ΕΦΣΑ του 2013 είχε προτείνει νέε δοκιμέ προκειμένου να προστατεύσουμε τι μέλισσε τόσο από τι αξίε όσο και από τι ε, χρόνε συνεπιστη τη έκθεση του σε αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Αλλά οι επιχειρήσει που τα κατασκευάζουν είχαν αντισταστεί σε αυτό και γνωρίζουμε ότι και στο Συμβούλιο υπήρξε μεγάλη αντίσταση ε, και το Συμβούλιο κάνει τώρα νέε αναθεωρημένε προτάσει προκειμένου να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Και η Επιτροπή αναφέρθηκε στο γεγονό ότι την λυπεί η κατάσταση όσο έχει σήμερα. Ε, θα ήθελα να μου επιβεβαιώσει η Επιτροπή ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο ε, ότι εάν ε, βγούμε από αυτό το αδιέξοδο και δεν υπάρξουν αντιρρήσει δηλαδή από την πλευρά των κρατών μελών θα είναι σε θέση η Επιτροπή να υποστηρίξει τα όσα είχαν υποστηριχθεί το 2013. Μάρτιν Όσλεγγ λέει τώρα. η Επιτροπή ε, λέει ότι οι προτάσει που κάνει τώρα αποτελούν βελτίωση, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι εσφαλμένο, γιατί μα λέει πω ε, η αξιολόγηση που κάνει τώρα αφορά μόνο τι οξύε επιπτώσει, αλλά όχι τι χρόνιε. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Ε, γιατί είχαμε κάνει και πολύ συγκεκριμένε, είχαμε διατυπώσει πολύ συγκεκριμένε αξιώσει γνωρίζουμε ότι μέλισσέ μα ε, πεθαίνουν, οπότε οι χρόνιε επιπτώσει, οι οποίε δυνητικά είναι πολύ πιο επικίνδυνε, τώρα δεν λαμβάνονται καν υπόψη. Γνωρίζουμε πώ εξαφανίζονται ακριβώ ε, σμήνοι ε, και δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την εξαφάνιση των μελισσών, γιατί το 84% και τη χλωρίδα εκεί που υπάρχουν βασίζεται στις μέλισσες και για τον ε, επικονιασμό τους. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι και η Επιτροπή αυτό που λέει ότι δηλαδή ελπίζει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα γίνει κάτι ε, περαιτέρω. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στα κράτη-μέλη ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Ε, δηλαδή ε, δεν επαρκεί ε, σε επίπεδο των όσων χρειαζόμαστε ως δεδομένα σε επιστημονικό επίπεδο και δεν ε, επαρκεί αυτό για να καλύψει και τις ανησυχίες του Εβραίου κοινού. Δηλαδή ουσιαστικά θα γελιοποιηθούμε αν πούμε ότι βασιζόμαστε σε αυτό. Για το ID τώρα, Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έθεσε αυτό το θέμα, το οποίο είναι τόσο λεπτό που συχνά όμως το παραβλέπουμε αδίκως. Όπως ποσοστά, πολύ σωστά είπατε, ε, υπάρχουν τεράστιες επιπτώσεις για τον πλανήτη μας και για την επισητιστική ασφάλεια οι μέλισσες. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια μόνιμη παρακολούθηση και να δημιουργήσουμε ομάδες εργασίας τεχνικές μόνιμες στα κράτη-μέλη που θα επιτρέψουν να ελέγξουμε την ε, υγεία των ε, μελισσών σε διάφορες περιοχές και σε διάφορα κλίματα και να υπο... υποβάλουμε προτάσεις για να προστατεύσουμε την υγεία τους και να τις υποβάλουμε στους α, ε, μελισσοκόμους και να τους αφυπνίσουμε σε σχέση με το πρόβλημα των ε, ε, προϊόντων φυτοπροστασίας. υπάρχουν α, οικολογικές πτυχές, θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη, τοξικολογικές και περιβαλλοντικές ε, και θα πρέπει η Κομισιόν να εξισορροπήσει τα διάφορα συμφέροντα, ε, να δει ε, τα συμφέροντα της χημικής βιομηχανίας, της γεωργίας και της μελισσοκομείας επίσης. Καθώς και το εθνικό βεβαίως και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Thank Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους ε, συναδελφούς για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας έκαναν. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το να διατηρήσουμε τους πληθυσμούς των ε, μελισσών μας ε, σε υγιή επίπεδα και γενικά των επικοινωνιστών μα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη διατήρηση των οικολογικών συστημάτων μας. Γι' αυτό το λόγο και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα. Πρώτον, πώς η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι τα φυτοφάρμακα δεν θα έχουν απαράδεκτες χρόνιες ή οξύες συνέπειες στην υγεία των μελισσών και των υπόλοιπων επικονιαστών με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Και δεύτερον, ε, πώ μπορούμε να εφαρμόσουμε πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, την αρχή τη προφύλαξη ε, όταν έχουμε δει ότι υπάρχει ακριβώ μια τέτοια ζημία, αλλά δεν έχουμε αντιμετωπίσει αυτέ τι συνέπειε εφόσον δηλαδή δεν έχουμε ζητήσει από τις αρμόδιες επιχειρήσεις να υποβάλουν τα δεδομένα που καταδεικνύουν ότι δεν έχουν βλαβερές συνέπειες όχι μόνο για τις μέλισσες αλλά και τους επικονιαστές. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος το ΕΛΚ και το ECR είχαν μείνει τώρα ως ε, πολιτικές ομάδες που δεν είχαν πάρει ακόμα το λόγο, οπότε για το ΕΛΚ και κυρία Νόβακ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και καλημέρα σε όλους. Πέρυσι, η 20η Μαΐου ανακηρύχθηκε ως η μέρα της Μέλισσας και η Σλοβενία ήταν η χώρα εκείνη η οποία είχε προτείνει ε, ε, ανακήρυξη αυτή τη ημέρα, ω ημέρα των μελισσών και έλαβε την υποστήριξη και άλλων κρατομέλων και μα χαροποιεί αυτό το γεγονό γιατί οι μελισσέ πραγματικά είναι πολύ σημαντικέ και για την ε, δική μα ζωή. Ότι δηλαδή είναι κακό για τις μέλισσες είναι αρνητικό και για μας, για τους ανθρώπους σε μακροπρόθεσμα. Ναι, χρειαζόμαστε φυτοπροστασία στον αγροτικό τομέα, αλλά δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε. Θα πρέπει να αξιώνουμε συνεχείς βελτιώσεις, δηλαδή προϊόντα τα οποία έχουν λιγότερες βλαβελές συνέπειες για τα ζώα, για τα, ε, τις αλλά και για τους ανθρώπους. Δεν θα πρέπει να υποκύπτουμε στις πιέσεις που ασκούν τα διάφορα λόμπι και η χημική βιομηχανία, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να ε, βρουν την εύκολη λύση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το θέλουμε εμεί. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, η κυρία Μάκιντάιρ τώρα για το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, και ζητώ συγγνώμη που κατέφθασα αργοπορημένη. Ελπίζω να μην θέσω λοιπόν ερωτήματα τα οποία ήδη έχουν απαντηθεί, αλλά θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα από πλευρά μου. Πρώτον, ε, πώ θα διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πω η αναθεωρημένη εκδοχή αυτού του εγγράφου καθοδήγηση ε, δεν θα βρει την ίδια αντίθεση από την πλευρά των κρατών μελών. Και ποια θα είναι η διαδικασία μόλις η ΕΦΣΑ ολοκληρώσει την επιστημονική της αξιολόγηση. Τα κράτη-μέλη θα έχουν συμμετάσχει, δηλαδή θα συμμετάχουν, συμμετέχουν και με συγκεκριμένε επιστημονικέ περιπτώσει. Δεύτερο τώρα ερώτημα. Ε, Προφανώ ε, χαιρετίζουμε το υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνη ε, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει η ΕΦΣΑ στο πλαίσιο αυτή τη αναθεώρηση, αλλά ήθελα να να ρωτήσω ποιε είναι οι άλλε δράσει που έχει αναλάβει προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άλλοι παράγοντε οι οποίοι επηρεάζουν την υγεία των μελισσών. Δηλαδή το γεγονό ότι αργοπεθαίνουν δεν έχουν αρκετή αρκετή χλωρίδα για να τραφούν, ο καταχαιρματισμός των σμηνών και ούτω καθεξής. Όλοι λοιπόν αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι έχουν αρνητικό αντίκτυπο ε, στους πληθυσμούς των μελισσών μας. Ε, εάν τους αγνοούμε αυτούς τους ε, παράγοντες εστιάζοντας μόνο στο ζήτημα των φωτοφαρμάκων, δεν βράθουμε σωστά. Ευχαριστώ, λέει ο για το ΕΛ και κυρία Σνάιντερ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήδη αναφέρθηκε ότι τον Απρίλιο του 2018 απαγορεύτηκαν τρία νέα νοικοτινοειδή, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την, ε, τις καλλιέργειες της αλλά στη συνέχεια υπήρξαν διαφορετικέ καταστάσει ό,τι αφορά την έγκριση αυτών των προϊόντων. Δηλαδή σε ορισμένα κράτη-μέλη υπήρξαν κάποιε ε, άδειε, οι οποίε τελικά χορηγήθηκαν ω άδειε έκτακτη ανάγκη. Ε, οπότε θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ακριβώς κάνει ε, σε σχέση με τέτοιου είδους εγκρίσεις έκτακτης ανάγκης και τι θέλει να κάνει στο μέλλον έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ομοιομορφία του κανονιστικού πλαισίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Για το Ρενιό, Φρέντερη Κρίς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πράγματι, πολλά χρόνια τώρα ζητάμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει πλήρη κριτήρια αξιολόγησης των επιπτώσεων ε, στις μέλισσες ε, και στην επικονίαση οι πολίτε είναι αυτοί που το ζητάνε, οι οποίοι απευθύνονται σε εμά κατά χιλιάδε. Μιλάω για του επιστήμονε, μιλάω για, του ίδιου του μελισσοκόμου. Ακόμα και για μα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη τον Ιανουάριο είχαμε την έκθεση τη ειδική επιτροπή μα για τα παρασιτοκτόνα, με τα φυτοφάρμακα συγγνώμη. Πολλοί συνάδελφοι υπέβαλαν πολύ συγκεκριμένε ε, τροπολογίε για το θέμα που συζητάμε σήμερα. Δεν μιλάω για τι χώρε μέλη, τα είπαν οι συνάδελφοι. Οπότε, τον αποφασιστεί μέσα στο καλοκαίρι νέα μέτρα αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη μόνο ένα κριτήριο, δηλαδή την άμεση έκθεση των μελισσών στις σχετικές ουσίες, αυτό νομίζω ότι αποκλίνει από αυτά που θέλουμε, γιατί δεν έχουμε υπόψη μας τις επιπτώσεις, τις νύμφες και άλλα. Τη... Μας είπε η Επιτροπή ότι πρόκειται για μέτρα που δείχνουν κάποια πρόοδο. Για μένα όχι. Οπισθοχωρούμε πιστεύω. Έχω μια ερώτηση με αυτό το κάτστιά ένα λεπτό δεν προλαβαίνουμε. Εδώ σε επιτροπέ δεν έχουμε αυτή τη συνήθεια. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να αναπτύσσουμε τα επιχειρήματά μας. Πρόεδρο, στόχο είναι να μπορέσουν περισσότεροι να υποβάλουν ερωτήσει. Και σε ένα λεπτό μπορεί κανείς να υποβάλει ερώτηση. Πράσινη. Μπάρι. Η κυρία Μπάρις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συμφωνήσω με τους συναδέρφους ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να τοποθετηθεί με στένος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσει να μην αφήσει τις χώρες μέλη να παραβιάζουν τον νόμο και τους κανόνες. Μετά από όλα αυτά που μας είπατε, πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι δεν θα αγνοείται η επιστημονική γνώση. Τώρα βασιζόμαστε στα επιστημονικά στοιχεία του 2002. Ακόμα και για την κλιματική αλλαγή λέμε ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τα επιστημονικά δεδομένα. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δυνατόν να αφήσει τις χώρες μέλη να κρύβονται πίσω από τα λόμπι. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ο κύριος Όρτσεκ από το Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύσκολα να μην επαναλάβει κανεί όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι με του οποίου συμφωνώ, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτή η Επιτροπή και ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει την αντίρρηση και να υποβάλει τελικά αυτή την ε, αντίρρηση. Και είναι κρίμα, ε, είναι ντροπή αυτό που κάνουν οι χώρε μέλη, που κρύβονται ουσιαστικά. Γιατί τελικά αυτό που έχουμε μπροστά μας εδώ είναι μια πρόταση η οποία παραβιάζει την νομοθεσία. Δεν κάνει τις αξιολογήσεις για, τις για τη χρόνια έκθεση και συνεπώς δεν τηρεί το γράμμα του νόμου. Αυτή η χρόνια έκθεση στην τοξικότητα είναι και το στοιχείο κλειδί. Άμα δεν ξέρουμε πώς να την αξιολογήσουμε, άμα δεν έχουμε συγκεκριμένη μεθοδολογία, πώς θα γίνει. Θα έπρεπε να υπάρχει. Εφόσον δεν υπάρχει μεθοδολογία, πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτές τις επιπτώσεις. Αλλά επίσης υπάρχει και ένα ενδιαφέρον επιχείρημα που ακούγεται για το πώς θα... Α, έληξε ο χρόνος μου. Καλά, συγγνώμη. Πρόεδρος, ωραία, ήδη έχουμε περάσει το χρόνο. Επιστρέφουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέντε λεπτά παρακαλώ να μας απαντήσετε ε, να απαντήσει σε ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε πέντε ερωτήσεις. Θα εστιάσω στις πιο σημαντικές, μερικές ίσως να τις παραβλέψω. Ε, κύριος Ντέιβις, ξεκινάμε αυτόν. Ε, η Κομισιόν υπέρ μιας πλήρους εφαρμογής. Ναι, είμαστε. Αυτή ήταν η αρχική μας πρόταση στη Μόνιμη Επιτροπή. Προτείναμε μόνιμη και πλήρη εφαρμογή της, ε, καθο, της κατεύθυνσης των κατευθυντήριων γραμμών. Επομένως, ναι είναι η απάντησή μου. Όπως ε, υπόθηκε πολύ σωστά, τα περισσότερα κράτη-μέλη απλώ ήταν αντίθετα. Όπως είπατε, κύριε Άικχορτ, δεν μπορούμε να κάνουμε μια πρόταση στο Συμβούλιο. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν οι κανόνε επιτροπολογία που απαιτούν να εξετάσουμε μια πρόταση που έχει τη μέγιστη στήριξη στην επιτροπολογία πριν κάνουμε την πρόταση στο Συμβούλιο. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε για συμβαστικέ λύσει. Συχνά συμβαίνει αυτό στι συζητήσει μα με τα κράτη-μέλη. Επίση, να τονίσω κάτι που είπαν πολλοί ευρωβουλευτέ, ότι πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ε, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε βελτιώσει. Συμφωνούμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Θα βελτιώσουμε ένα τμήμα τη ε, αξιολόγηση του κινδύνου, όχι τα πάντα, το ξέρουμε. Γιατί δεν μα αφήνουν τα κράτη-μέλη να βελτιώσουμε τα πάντα σε αυτή τη φάση κυρία Ακχούλ. Δεν αποδυναμώνουμε τα πρότυπα. Δεν συμφωνώ με αυτό. Ε, το παράδειγμα με τα νέο νεονικοτινοειδή που χρησιμοποίησατε και είπατε ότι θα οδηγήσει σε διπλά πρότυπα. Όχι. Κάνουμε αυτή την έκτακτη αναθεώρηση ε, για τα νέο νεονικοτινοειδή. Η αρχική έγκριση βασίζονταν στις, στα πρότυπα του 2002. Μετά τα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ ζητήσαμε από τις εταιρείες να να υποβάλουν επιπλέον ε, δεδομένα που αξιολογούνται με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές. Ε, κυρία Γκούτελα. Ναι, ζητάμε από την ΕΦΣΑ να χρησιμοποιήσει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές στα συμπεράσματα. Ε, σε ό,τι αφορά την νομική απόφαση, είμαστε υποχρεωμένοι όμως να εφαρμόσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του 2002, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια έγκαιρη αναθεώρηση όταν δούμε τα προβλήματα και να χρησιμοποιήσουμε τις νέες ε, την αναθεώρηση, όπως επιβεβαιώθηκε από το δικαστήριο. βεβαίω, αυτή η απόφαση έχει προσβληθεί τώρα. Έχει γίνει προσφυγή εναντίον τη. Θα πρέπει να δούμε πώς θα τελεσυνδικήσει. Ε, κύριε Χόστινγκ, δεν κάνουμε ένα βήμα προ τα πίσω, δεν υπάρχει αναχώρηση. Αντίθετα, αν ο κανονισμός που προτείνουμε σήμερα δεν υιοθετηθεί, τότε παραμένουμε σε αδιέξοδο εκεί που έχουμε μείνει τα επόμενα πέντε ε, χρόνια αν, δεν, ε, αν υιοθετηθεί, θα γίνει ένα βήμα προς τα εμπρός. Δεν είναι το 100% αλλά κάτι είναι. Και να επανέλθω στο ερώτημα του αν θέλουμε πιστεύουμε ότι οι νέε κατευθυντήριε γραμμέ τη ΕΦΣΑ μετά την αναθεώρηση θα υιοθετηθούν. Ναι, θα υιοθετηθούν. Γιατί ζητήσαμε από την ΕΦΣΑ να εμπλέξει τα κράτη-μέλη και τους εμπειρογνώμονες από τους άλλους stakeholders σε όλη τη διαδικασία. Ήταν ένα από τα στοιχεία ούτω ή άλλω που οδήγησαν στην απόρριψη των κρατών μελών. Το γεγονό ότι δεν εμπλακήκαν ή έτσι πιστεύανε στη διαδικασία που οδήγησε στι κατευθύνσει γραμμέ του 2013. Είναι δική του πεποίθηση. Και εμεί και η ΕΦΣΑ δεν συμφωνούμε. Εμεί πιστεύουμε ότι το εμπλέξαμε, αλλά αυτό ισχυρίζονται. Γι' αυτό δεν υποστήριξαν την πλήρη εφαρμογή. Είμαστε δεσμευμένοι τώρα να το περάσουμε αυτό, να κάνουμε βελτιώσεις και θα θέλαμε και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να μας ε, στηρίξει για να κάνουμε αυτό το μερικό βήμα προς τα εμπρός, παρότι δεν είναι το 100%. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε πλήρως. Ευχαριστώ που δεν χρησιμοποίησατε και το πεντάλεπτο λόγο και ήσασταν τόσο ακριβείς. Είναι μια πρώτη συζήτηση αυτή. Η επόμενη θα γίνει αφορά την ε, προθεσμία ε, για την αντίρρηση που είναι μέχρι την ε, Παρασκευή. Και θα επανέλθουμε σε ψηφοφορία εδώ και αν χρειαστεί και στην Ολομέλεια. Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη συζήτηση με την Κομισιόν και πάμε στην ανταλλαγή απόψεων με την ΕΦΣΑ. Πού είναι ο πρόσωπος της ΕΦΣΑ? 10 λεπτά έχετε για 10 λεπτά έχετε το λόγο. Είσαστε ε, τμηματάρχης της μονάδας φυτοφαρμάκων ή τμηματάρχης. Οι συζητήσεις έχουν σχέση αυτές οι δύο συζητήσεις. Η παρουσίασή σας όμως αφορά το ίδιο το έγγραφο και αν έχετε υπόλοιποι ερωτήσεις Μπορείτε βεβαίω να χρησιμοποιήσετε και τα όσα υπόθηκαν στην προηγούμενη συζήτηση, αλλά α ξεκινήσετε εσεί εύσα με την παρουσίαση του εγγράφου σα. Δέκα λεπτά. Μανουέλα Τιραμάνη λέγομαι. Θέλω να τα βασικά. Θέλω να ξεκινήσουμε το, τα βασικά στοιχεία του εγγράφου του 2013. Τότε οι εμπειρογνώμονες που είχαν εμπλακεί στη δουλειά είχαν εντοπίσει ότι κάθε, κάθε κάποιοι τομείς για την αξιολόγηση δεν είχαν ληφθεί υπόψη. Κάποιοι κανόνες έκθεσης, ας πούμε. Ο στόχος των κατηγοριών γραμμών του 2013 ήταν να καλυφθούν κάποια κενά και να έχουμε και συστήματα για τις αγριομέλισσες και τις μεμονωμένες μέλισσες όχι μόνο για τις μέλισσες των ε, σμηνών και κυψελών. Μια νέα μεθοδολογία επίσης ε, χρησιμοποιήθηκε για να δούμε εάν ένας κίνδυνος, να αποφασίσουμε ένας κίνδυνος είναι αποδεκτός ή όχι. Ο στόχος του εγγράφου ήταν να φτάσουμε σε ένα εργαλείο για τους ε, stakeholders, τους ενδιαφερόμενους φορείς και φυσικά τα κράτη-μέλη, τις δημόσιες αρχές και το κλάδο, ούτω ώστε να, δώσουν, να δώσει δεδομένα για να κάνουν σωστή αξιολόγηση του κινδύνου. Η προσέγγιση μας ήταν διτή. Ξεκινούσε από ένα πρώτο επίπεδο, ένα απλό πρώτο επίπεδο και προχωρούσαμε ανάλογα με το αποτέλεσμα σε πιο ε, λεπτομερή αξιολόγηση κινδύνου, πιο περίπλοκη βεβαίως, γιατί θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε και μελέτες και επιτόπιες μελέτες. Όπως είπα και ο Κλάους πριν από μένα, κάποιες καινοτομίε για την έκθεση, παραδείγματο χάρη ε, κατά κάποια ε, ψεκασμών, ε, νερό κτλ, ε, πηγές έκθεσης, παραδείγματο χάρη λουλούδια, ε, ζυζάνια και άλλα πράγματα. Επίσης, ε, λάβαμε υπόψη μας ε, την έκθεση στους μεταβολίτες ε, που υπάρχει στο νέκταρ των επικονιαστών και που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι μέλισσες. Βασικό στοιχείο της δραστηριότητας τότε, που ισχύει και τώρα, ήταν να καθορίσουμε, ε, να ορίσουμε κάποιους ε, στόχους προστασίας που καθορίστηκαν με διαβούλευση, έντονη διαβούλευση, με τους ε, διαχειριστές του κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε τι είναι όλο αυτό. Ο ορισμός του μέγιστου επιτρεπτού επίπεδου ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στις μέλισσες χωρίς να έχει αρνητική επίπτωση στις υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Δηλαδή, είναι οι δραστηριότητες αυτές, αυτές οι υπηρεσίες, που, κάνουν, που προσφέρουν και κάνουν οι μέλισσες, που είναι ο ε, επικονιασμός. Αυτός ο ορισμός προέκυψε ε, με κάποια χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας υπόψη κάποια χαρακτηριστικά πρέπει να προστατεύσουμε. Παραδείγματος χάρη, η επιβίωση, ανάπτυξη των απικιών, πολλοί από εσά αναφέρατε και την υγεία των, α, της, της κάμπιας. Πρόσφατα ε, λάβαμε την εντολή να αναθεωρήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές γιατί η πλειοψηφία των κρατών μελών δεν τα ενέκριναν και ζήτησαν επικαιροποίηση με βάση νέα επιστημονικά στοιχεία τα οποία έχουμε πλέον τώρα, αφού πέρασαν κάποια χρόνια. Η αναθεώρηση εστίασε κυρίως, αλλά όχι μόνο, ε, στην έννοια της εθνισιμότητας της μέλισσας ε, και λαμβάνοντας ε, ρεαλιστικά στοιχεία διαχείρισης της μελισσοκομείας και τη φυσική εθνισιμότητα. Δρόμους έκθεσης, επίσης, οδή έκθεσης, που έπρεπε να ληφθούν υπόψη και κυρίως η έκθεση από δραστηριότητες ε, ψεκασμού ή τι γίνεται με την, ε, όταν χρησιμοποιούμε φυτο, προϊόντα φυτοπροστασίας για τους πόρους κτλ. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ε, ποιες καλλιέργειες ελκύουν τις ε, μέλισσες. Ε, η μεθοδολογία αυτή είναι σημαντική ειδικά για το πιο ε, περίπλοκο επίπεδο. Εκεί θέλουμε επιπλέον πληροφορίες. Ε, επίσης υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ε, ένα σχέδιο εργασίας, όλοι μπορείτε να το δείτε. Θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά το Μάρτιο του 2021 και φυσικά εξαρτόμαστε ε, από τους ορισμούς των διαχειριστών του κινδύνου για τους στόχους. Ε, είναι σημαντική η εμπλοκή των ε, διαφερωμένων φορέων. Ε, για αυτές τις κατευθυντικές γραμμές συνεργαστήκαμε πολύ από την, τους συναδέλφους, με τους συναδέλφους και με τους stakeholders. Το σχέδιο εδώ δεν το βλέπετε καλά. Θα το συνοψίσω. Υπάρχουν διάφορα βήματα διαβούλευσης. Τη δουλειά που κάνουμε εμείς εσωτερικά, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, τα πρωτόκολλα για το πώς θα ορίσουμε και πώς θα συλλέξουμε και θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα για την θνησιμότητα και συνεχεία δημόσια διαβούλευση των, των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών. Ένα εργαστήρι θα γίνει επίσης για να συζητήσουμε με τους stakeholders απευθείας τα σχόλια που λάβαμε και συνεχεία θα υπάρξει η οριστικοποίηση. Ε, δεσμευόμαστε να κάνουμε διάφορα επίπεδα παρουσίασης και συλλογής ε, αντιδράσεων στην ε, Επιτροπή και στο δίκτυο φυτο, προϊόντων φυτοπροστασίας που έχει η ΕΦΣΑ με συναδέλφους από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Thank you very much. So the presentation... Σας ευχαριστώ. αυτή η παρουσίαση θα διανεμηθεί στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να έχει πρόσβαση. Ε, σε έντυπη μορφή σε αυτό το έγγραφο κιόλας. Τώρα θα κλείσω ο κατάλογος των ομιλητών ε, που θέλουν να πάρουν το λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας Catch the Eye. Αν υπάρχει κάποιος ακόμα στη τώρα. Καλώς λοιπόν, θα ξεκινήσω από την ΚΟΕ γιατί ε, αυτή ήταν η πολιτική ομάδα που έκανε πρώτη την πρόταση να έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα εδώ ε, με την ΕΦΣΑ, οπότε δίνω το λόγο στην κυρία Χάζακα εκ μέρους της Γουέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εδώ και πολλά χρόνια ανεξάρτητοι επιστήμονες ε, μας προειδοποιούν σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα, ειδικότερα ε, τα νέο νοικοτινοειδή για τις μέλισσες. Αλλά ακόμα δεν έχουμε ε, δημιουργήσει τα απαραίτητα επιστημονικά μοντέλα προκειμένου να αποκλείσουμε από τις διαδικασίες έγκρισης αυτά τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα. Οι κατευθυντήρε γραμμές για τις μέλισσες της ΕΦΣΑ του 2013 έχει δεχθεί ισχυρά πειρά από τα λόμπι της χημικής βιομηχανίας και ουσιαστικά αυτό το έγγραφο έχει τεθεί εκτός ε, εφαρμογής από το Συμβούλιο, επειδή ακριβώς το Συμβούλιο έχει υποκύψει στα συμφέροντα της χημικής βιομηχανίας και κατά συνέπεια ακόμα και σήμερα επιτρέπονται αυτά τα προϊόντα στην αγορά. Σας ε, ρωτώ λοιπόν, Πώ αυτή η διαδικασία διαβούλευση που έχετε κινήσει τώρα θα μα οδηγήσει σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε δηλαδή ότι στην ομάδα των stakeholders, των ενδιαφερομένων φορέων, έχουμε υπερεκπροσώπηση από την πλευρά των λόμπι και γνωρίζουμε πω αυτοί οι παίκτε ε, έχουν πολύ χρόνο και χρήμα στη διάθεσή του έτσι ώστε να κάνουν ό,τι μπορούν ε, προκειμένου να λάβουν τι άδειε που θέλουν και να μην περιοριστεί η πρόσβασή του στην αγορά. Και βλέπουμε κράτη-μέλη ε, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τι κατευθυντήριε γραμμέ σα. Οπότε πώ τι θα κάνετε για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν νομίζω πως η διαμάχη αυτή θα επιληθεί ε, μέσω ομάδων διαβούλευσης, οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι της χημικής βιομηχανίας. Όχι, θα χρειαστούμε επιστημονικά δεδομένα και η μόνη, αν θέλετε, ενδιαφερόμενη φορείς είναι οι μέλισσες, οι πεταλούδες και άλλα έντομα. Και γνωρίζετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτά τα έντομα. Και δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε οικονομικού χαρακτήρα επιχειρήματα για να επιλύσουμε μια οικολογικού χαρακτήρα λύση. Και θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Ε, το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το ποια μοντέλα θα πρέπει να εφαρμόσουμε ώστε να περιορίσουμε τη θνησιμότητα των μελισσών και το πώ θα κάνουμε επιτόπιε μελέτε. Οπότε, ποια είναι η άποψη τη ΕΦΣΑ και γιατί δεν επιθυμεί τέτοιου είδου μελέτε ο κλάδο. Και δεύτερο ερώτημα. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ε, ο, τα επίπεδα των αποδεκτών απολειών δεν θα πρέπει να μετρούνται σε αγροτικό επίπεδο αφού ήδη οι, ε, τα, αυτές οι αγροτικές περιοχές είναι ήδη μολυσμένες με ε, φυτοφάρμακα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Έχω έξι ακόμα συναδελφούς που έχουν στήσει το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στον καθένα από αυτούς για 1,5 λεπτό. Η κυρία Κόβαξ ε, τώρα εκ μέρους του ΕΛΚ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. από το 2015 και μετά όλοι οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δεδομένα ε, σε σχέση ακριβώς με την τοξικότητα ή μη των προϊόντων τους. Ωστόσο δεν έχουμε κάποιους ε, τρόπους για να επαληθεύουμε αυτά τα δεδομένα. Ε, ποια είναι λοιπόν η δική σας αξιολόγηση. Πράγματι επιρρούν αυτές τις υποχρεώσεις τους οι παραγωγοί σε ό,τι αφορά την χορήγηση δεδομένων σε σχέση με την τοξικότητα των προϊόντων τους ή αντιθέτως θεωρείτε ότι υπάρχει έλλειψη σε ό,τι αφορά τα παρεχόμενα δεδομένα. Επίση, τα εν λόγω δεδομένα θεωρείται πω είναι επαρκή, έχουν το απαραίτητο επίπεδο ποιότητα και τι μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει κάποιο σίγουρο τρόπο για να αξιολογήσουμε τη σήμερα ημέρα την ταξικότητα ε, κάποιων τέτοιων προϊόντων. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές τώρα, κυρία Πόζακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάτι προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει, εμείς είχαμε αναφερθεί στο έγγραφο της καθοδήγησης ε, για τις μέλησες ε, και το γεγονός ότι πολλές κυβερνήσεις ε, κρατών μελών δεν έχουν εφαρμόσει την εν λόγω καθοδήγηση, ενώ κάποιες από αυτές τις κυβερνήσεις είχαν αντιταχθεί σε αυτή η ανησυχία μου τώρα είναι ότι οι ίδιοι αξιωματούχοι από τι ίδιε κυβερνήσει είναι εκείνοι που συμμετέχουν στη διαδικασία αναθεώρηση του ίδιου εγγράφου καθοδήγηση. Διαρωτώ με λοιπόν, πώ η ΕΦΣΑ θα διασφαλίσει ε, την παροχή συμβουλών στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία διαβούλευση ε, που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και θα είναι αξιόπιστη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, ε, για το Renew τώρα, ο Chris Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε λοιπόν από την Επιτροπή να μα λέει ότι υποστηρίζει ε, την καθοδήγησή τη ΕΦΣΑ το 2013, καθοδήγηση η οποία έχει μπλοκαριστεί από το Συμβούλιο. Και γνωρίζουμε ότι τώρα έχει ζητηθεί από την ΕΦΣΑ να προβεί σε μια διαδικασία αναθεώρηση του ελογόγραφου. Οπότε, ερωτώ τον πρόσωπο τη ΕΦΣΑ δύο ε, τεινά. Πρώτον, εσεί εσείς υποστηρίζετε τα επιστημονικά δεδομένα αυτών των συμπερασμάτων της αξιολόγησης του 2013 και τι θεωρείτε εσείς, ποιες θεωρείτε πως θα είναι επιπτώσεις για τις μέλισσες και τους επικονιαστές εάν τελικά το αποτέλεσμα αυτής της αναθεώρησης ε, θα είναι ένα αποδυναμωμένο νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων σε σύγκριση με εκείνο του 2013. Πάει σε τώρα για τους πράσινου. παρακαλώ. Σας ευχαριστώ ουσιαστικά αναφερόμαστε στα ίδια ερωτήματα, αλλά τελικά εσείς ΕΦΣΑ δημιουργήσατε, καταρτήσατε αυτό το έγγραφο καθοδήγησης του 2013, αλλά τα κράτη-μέλη είπαν ότι είναι υπερβολικά συντηρητικό αυτό το έγγραφο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Και μάλιστα αυτή η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη είναι η ίδια με αυτή που, χρησιμοποιούν, ε, χρησιμοποιεί ο κλάδος. Ε, μάλλον είναι σύμπτωση άλλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, εσείς, κατά τη δική σας άποψη, κατά την άποψη ΕΦΣΑ, θεωρείτε πως θα πρέπει πράγματι να γίνει αναθεώρηση αυτή τη ε, καθοδήγηση ή σα ε, πίεσαν τα κράτη-μέλη να το πράξετε. Και επίση, πώ θα διασφαλίσετε ότι στο πλαίσιο αυτή τη αναθεώρηση τα επιστημονικά δεδομένα θα είναι και υψηλή ποιότητα αλλά και αμερόληπτα, από αμερόληπτε πηγέ. Γιατί έχω την αίσθηση ότι εσεί ουσιαστικά εμ, εμ, είστε υποχρεωμένοι τώρα ως ΕΦΣΑ να προβείτε και στη διαχείριση των κινδύνων αλλά και στην αξιολόγηση των κινδύνων ταυτόχρονα που είναι δύο ξεχωριστά. Οπότε ε, σας ερωτώ, θεωρείτε πως ε, το έγγραφο καθοδήγησης που είχατε κατατήσει το 2013 ήταν ελλειπές. Ευχαριστώ για το ΕΛΚ, κυρία Νόβακ. So, ε, uh, Mr. Panie Przewodniczący, Παρακαλώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι ότι η ΕΦΣΑ είναι υπεύθυνη για την επιστημονική αξιολόγηση διαφόρων προϊόντων, όπως είναι τα φυτοφάρμακα, τα, μη, τα γενετικά τοπιμεμένα προϊόντα κλπ. κλπ. Αλλά είναι και υπεύθυνη για την εκπόνηση μεθοδολογίας, η οποία βοηθάει στην αξιολόγηση αυτή. Διαβάζοντας την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2018, εκπρόσωποι των Υπουργείων το μόνο που κάνουν είναι ότι υπογράφουν ε, τη μεθοδολογία για τα φυτοφάρμακα, αλλά όχι για άλλα προϊόντα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Εδώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει πραγματικά διάκριση ανάμεσα στη διαχείριση κινδύνου και την αξιολόγηση κινδύνου. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει. Η τελευταία κυρία Ριβαζή, εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε συχνά τα βάζουμε με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Εγώ ευχαριστώ την ΕΦΣΑ, δεν το κάνω κάθε μέρα, γιατί οι κατευθυντήριες γραμμές του 2013 ήταν καλές, έγκυρες, γιατί λαμβάνουν υπόψη και τις οξύες επιπτώσεις και τις χρόνιες, αλλά και τις πηγές ρήπανσης. Αν λοιπόν πρέπει να επικρίνει κανείς κάποιον, είναι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι χώρε μέλη. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2018 ήταν ειλικρινή, γιατί είχε συνεισφέρει για να απαγορευτούν τα νέο νοικοτινοειδή. Η χημική βιομηχανία, όμως και διάφορες κυβερνήσεις θέλησαν να αλλάξουν τα πράγματα. Οπότε η ερώτηση προς την ΕΣΦΑ είναι εξής. Ποια είναι η γνώμη σας για την αναθεώρηση, αφού εργαστήκατε επιστημονικά για την αξιολόγηση κινδύνων και υπήρξε και η Επιτροπή Φυτοφαρμάκων που είπε ότι πρέπει να συμπεριλάβουν περισσότερα πράγματα, ότι η ιστορία των επικονιστών είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη διατροφή. Ε, λοιπόν, ποια είναι η δικιά σας θέση για αυτά. Τι πιστεύετε για την ποιότητα των μελετών των κατασκευαστών, γιατί αυτοί κάνουν τις εκθέσεις, είναι ποιότητας όσον αφορά την ε, χρόνια τοξικότητα για παράδειγμα. Τρίτον, γιατί και με τι επιχείρημα η βιομηχανία έπεισε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη ότι έπρεπε να υπάρξει αναθεώρηση της οδηγίας, των επιστημονικών δεδομένων δηλαδή που εσείς είχατε εκπονήσει. Με τι κριτήρια, τι τους ενοχλεί περισσότερο. Και τέλος, για το ρυθμιστικό τμήμα. Εγώ πιστεύω ότι εδώ υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στον κανονισμό αυτό και τον 1107 που ζητάει να γίνονται μελέτες για τις χρόνιες επιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ακούσω την άποψή σας. Μην αλλάξετε. Σας λένε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί. Ε, πείτε κι εσείς πρέπει. Τι λέτε. Αν δεν το πιστεύετε, πείτε το. Πρόεδρος, ωραία. Θα δώσουμε το λόγο πάλι στην Εύσα. Για πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από την πρώτη ερώτηση για το πώς ε, υπάρχει εγγύηση ότι θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα αυτή τη φορά. Κοιτάξτε, εμεί βασιζόμαστε στην επιστήμη και την ποιότητα της επιστημονικής γνώσης. Αυτό είναι ο κύριος στόχος του έργου μας. Βασιζόμαστε πολύ βέβαια στη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων πλευρών κατά τη διαδικασία. Και οφείλω να πω, το είπαν και κάποιοι από εσά, ότι οι χώρες μέλη, κυρίως εκείνες που ήταν κατά των κατευθυντηρίων γραμμών, βάριναν. Εμείς όμως την ε, επιστήμη λαμβάνουμε υπόψη μας. Συμμετέχουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν την τεχνική γνώση και όχι αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται το θέμα. Τώρα για την παρουσία επιχειρήσεων. Έχουμε μια λεπτομερή διαδικασία στην ΕΦΣΑ για το ποιοι συμμετέχουν. Είναι μια προσέγγιση που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και έχουμε πολύ συγκεκριμένους κανόνες για το πώς συμμετέχει ο κόσμος, ποιοι εκπρόσωποι κτλ. Ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες και τους έχουμε χρησιμοποιήσει και σε πολλά άλλα πλαίσια τους ίδιους κανόνες και για άλλα έγγραφα. Ο στόχος μας τώρα είναι η επιστημονική πτυχή και οτιδήποτε άλλο είναι πέρα από τις δικές μας αρμοδιότητες. Τώρα για το θέμα της μεθοδολογίας. Θα έλεγα ότι εγώ δεν έχω προσωπική άποψη γιατί βασίζομαι σε επιστημονικά δεδομένα. Οπότε και γι' αυτό θα εξετάσουμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Και μετά τα δεδομένα αυτά θα τα παρουσιάσουμε στους συνεδέρφους που έχουν την ευθύνη να καθορίσουν τους στόχους προστασίας. Σε σχέση τώρα με την ποιότητα των μελετών που μας στάνουν από τους παραγωγούς είναι όπως και σε οποιαδήποτε άλλη αξιολόγηση κινδύνου που κάνουμε. Πάντα ελέγχουμε την ποιότητα των δεδομένων και ανάλογα με την ποιότητα αυτή αποφασίζουμε. Οπότε Κάθε μελέτη εξετάζεται βάσει του κριτηρίου της ποιότητας και έτσι λαμβάνεται υπόψη στη συνέχεια στην αξιολόγηση. Έτσι διασφαλίζουμε την ποιότητα, πλήρης ποιότητα. Όσον αφορά την ανεξαρτησία, ξέρετε ότι έχουμε μια ομάδα εργασίας η οποία ακριβώς αυτή τη δουλειά κάνει εξετάζετε, δηλαδή για την εξαρτησία όλες ε, τις ε, μελέτες Και, λοιπά και εξετάζεται και σύγκρουση συμφερόντων εφόσον υπάρχει. Εξετάζεται δηλαδή και αυτό το κριτήριο ενδελεχώς. Τώρα για το κατά πόσο στηρίζουμε τα επιστημονικά δεδομένα, ε, κοίταξτε σήμερα κοιτάμε τις εξελίξεις από το 2013 και θα δούμε κατά πόσο θα επηρεαστεί κάποια παράμετρο ή όχι. Δεν μπορώ αυτό να το προβλέψω τώρα, γιατί τώρα θα αρχίσει μόλι η εργασία αυτή την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, κατά πόσο πιστεύουμε ότι χρειάζεται αναθεώρηση. Όπως είπα, η επιστήμη μας καθοδηγεί, η επιστημονική γνώση. Στην επιστήμη 10 χρόνια είναι μεγάλη χρονική περίοδος. Θα δούμε λοιπόν ότι θα έχουμε μετά την ανάλυση όπως και σε άλλα πλαίσια, έτσι και εδώ, για κάποια καυτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, λίγα χρόνια φτάνουν για να υπάρξουν πάρα πολλές δημοσιεύσεις. Οπότε θα δούμε αν έχουμε νέα στοιχεία, ποια θα είναι τα ευρήματα. Όσον αφορά ε, τη σύνδεση της αξιολόγησης κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνου, δεν ξέρω αν ε, μπορώ να σας απαντήσω πλήρως, αλλά είναι μια συζήτηση που κάνουμε με τους συναδέρφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι τα κρατάμε διακριτά αυτά τα δύο στοιχεία. Ε, πραγματικά, σταματάμε στην αξιολόγηση κινδύνου και παρουσιάζουμε τα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Και γι' αυτό ζητάμε από τους ε, διαχειριστές να μας πούν τη γνώμη τους για τους στόχους προστασίας. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της ΕΦΣΑ για την πρόσκληση αυτή. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Τώρα, κλείνουμε αυτό το θέμα, την ανταλλαγή απόψεων δηλαδή με την ΕΦΣΑ όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις μέλισσες. Και περνάμε σε επόμενο θέμα στο δεύτερο τμήμα δηλαδή του σημερινού πρωινού με το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη και 7. Εδώ υπάρχουν πολλοί νέοι ευρωβουλευτές και η επιτροπολογία μπορεί να είναι δύσκολο θέμα για αυτούς. Θα σας εξηγήσω απλώ ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία συζήτησης, μιας αντίρρησης όσον αφορά εκτελεστικό ε, κανόνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην ημερήσια διάταξη έχετε όλο τον κατάλογο των προϊόντων που αφορούν οι αντιρρήσεις αυτές, δεν σας το διαβάσω. Και θα οργανώσουμε την συζήτηση ως εξής. Μαζί οι αντιρρήσεις 6 και 7, καταρχήν, γιατί πρόκειται για αντίρρηση που έχουμε από την ΚΟΕ. Η ΚΟΕ έχουν τον εισηγητή. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην ΚΟΕ για τέσσερα λεπτά για τις δύο αυτές αντιρρήσεις, σημεία 6 και 7. Όπως είπα, υπάρχουν πολλοί νέοι ευρωβουλευτές εδώ, οπότε ό,τι έχετε να μας πείτε για την διαδικασία και τα λοιπά, ευχαρίστως. Λοιπόν, για τέσσερα λεπτά η συγγήτρια, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Οι αντιρρήσεις δεν αφορούν όλες τις ουσίες που λέει ο τίτλος, κυρίως δύο. Το χλώρο των λωρών και την φλούμιο ξαζίνη. Να σας δώσω κάποιες γενικές πληροφορίες. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λέει ότι η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον θα πρέπει να προστατεύονται πάντα και τα οικονομικά συμφέροντα δεν θα πρέπει ποτέ να πριτανεύουν σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι με την αναθεώρηση της ε, χρήσης αυτών των ε, φυτοφαρμάκων γίνεται. Τοξίνε, ε, το, τοξικά προϊόντα υπάρχουν επί πολλά χρόνια στην ευρωπαϊκή αγορά μετά την εκπνοή της έγκρισής τους. Έχω αντίρρηση λοιπόν στην παράταση της ε, περίοδου έγκρισης για την ε, φλουμιοξαζίνη και την άλλη Η φλουμιοξαζίνη είναι τοξική για την αναπαραγωγική δραστηριότητα και είναι γνωστός ενδοκρινικός διαταράκτης. Το χλωροτολερόν είναι επίσης ε, ενδοκρινικός διαταράκτης και δημιουργεί πρόβλημα στο αγέννητο παιδί. Είναι τοξικά για την υδρόβια ζωή με μακρές συνέπειες και αυτό επιβεβαιώνει, το επιβεβαιώνει η ΕΦΣΑ και η ΕΚΑ και υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εδώ και τέσσερα χρόνια τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει στην ανάκληση της έγκρισης από την Κομισιόν εδώ και χρόνια. Το άρθρο 21 στον κανονισμό των φυτοφαρμάκων το επιβάλλει αυτό. Αντίθετα, χρησιμοποιούν το άρθρο 17 και παρατείνουν την έγκριση και το έχουν κάνει μάλιστα έξι φορές συναπτές. Αυτό αποδεικνύει ότι φοβάται η Κομισιόν την πολύ δυνατή χημική βιομηχανία, ότι θα τη μηνύσει και θα έλεγα στην Κομισιόν ας τολμήσουν. Δηλαδή, το περιβάλλον μας, η δημόσια υγεία ε, δεν έρχεται πρώτη. Ας τους αντιμετωπίσετε, ας αντιμετωπίσετε τη χημική βιομηχανία στο δικαστήριο. Γιατί έχετε τα επιστημονικά στοιχεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το νόμο το μέρος σας. Εάν τελικά αποφασίσετε να αντισταθείτε στην χημική βιομηχανία. Ε, η χρήση αυτών των ε, ουσιών είναι σε αντίθεση με τον κανονισμό των φυντοφαρμάκων. Ε, μόνο ε, οι ουσίες οι οποίες θεωρούνται ασφαλείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και είναι και αντίθετες αυτές οι ουσίες με την αρχή της πρόληψης της ε, συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποχρεώνει την Κομισιόν να προστατεύσει το περιβάλλον και την υγεία μας. Κομισιόν, μην επιτρέπετε αυτές τις επιβλαβείς ουσίες ε, στους κάμπους και στο πιάτο μας και ε, να αποσύρετε παρακαλώ αυτές τις δύο ουσίες από, από τον κατάλογο των ουσιών που εξαιρούνται. Θα πάρουν το λόγο οι σκιώδεις τώρα για την κοινή συζήτηση των 6 και 7. Θα ξεκινήσω με το ΕΛΚ. Τρία λεπτά ανά Αν έχετε δύο σκιώδεις συζητητές, ένα για το 6 και ένα για το 7, να μοιράσετε το χρόνο. 1,5 και 1,5 έκαστος. Αν έχετε έναν μομιλητή, έχετε τρία λεπτά η ομάδα. Η κάθε ομάδα έχει πάντως τρία λεφτά και στη διαχειριστεί όπως θέλει. Το ΕΛΚ έχει δύο σκιώδεις συζητητές. Κρίστιν Σνάιντερ και Μισελ Βιζίκ Μοιράστε τα τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Μπορώ να κατανοήσω πολύ καλά το σκεπτικό της εισηγήτριας και της ε, ατηρήσεις ε, που έχει σε ό,τι αφορά καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα τέτοια προϊόντα. Η χρήση τους δηλαδή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ περιορισμένη ή απαγορευμένη ή τουλάχιστον θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να αποκλεί κάθε είδους ευλαβερές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Άρα λοιπόν υποστηρίζω ε, την αξίωση που είχαμε κάνει και στο ψήφισμα το περσινό από τη δική μας πλευρά αλλά και στο πλαίσιο της ειδική Επιτροπής για τα φυτοφάρμακα ότι δηλαδή πάντοτε χρειαζόμαστε επιστημονικά δεδομένα και επιστημονική τεκμηρίωση για τη χρήση τέτοιων προϊόντων και θα πρέπει ε, ε, θεωρώ να ε, βελτιώσουμε και να εναρμονίσουμε πανευρωπαϊκά την σχετική νομοθεσία. Βέβαια αυτό δεν είναι το ζητούμενο σήμερα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο αυτές οι 34 ουσίες θα παραταθούν σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις που έχουν ή όχι για διάθεση στην αγορά κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να μην ανανεωθούν ή να ανακληθούν οι εν λόγω άδειε. Σε ό,τι αφορά την εν λόγω διαδικασία, οι νόμοι εδώ είναι πολύ ξεκάθαροι, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν οι αξιολογήσεις δεν έχουν γίνει εγκαίρως, τότε και η σχετική καθυστέρηση δεν αποτελεί πετιότητα του ε, κατασκευαστή, τότε ε, είναι υποχρεωμένη να παρατείνει την άδεια. Ε, και πράγματι αυτό ισχύει σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή η αξιολόγηση από την πλευρά των αρχών αξιολόγηση των κρατών μελών είναι που έχει καθυστερήσει και όχι από την πλευρά των επιχειρήσεων έχει λάβει χώρα αυτή η καθυστέρηση και αυτό βέβαια ήταν από τα κυριότερα σημεία κριτικής που άσκησε στο ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι. Άρα λοιπόν, ε, συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό, ότι η παράταση των αδειών ε, σε ό,τι αφορά αυτέ τι ουσίε, η σχετική απόφαση θα ληφθεί εντό τριών ή έξι μηνών. Εάν ακολουθήσουμε ε, βέβαια τις, όλες τις προτάσεις που κάνει η συγγήτρια, βεβαια τις ολες τις προτασεις που κανει η συγγητρια αυτο θα είχε πολύ μεγάλε συνέπειε, γιατί ουσιαστικά ε, με βάση μια αυθαίρετη απόφαση μια σειρά από ουσίε. δεν θα ήταν δυνατόν πλέον να κυκλοφορούν, χωρί όμω αυτό να έχει βασιστεί σε επιστημονικά δεδομένα. Ε, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θα υπονομεύσουμε ε, και τη δυνατότητα σχεδιασμού μακροπρόθεσμα από την πλευρά των γεωργών μα. Αλλά αυτοί χρειάζονται μια τέτοια δυνατότητα γιατί ακριβώ βασίζονται στη χρήση αυτών των προϊόντων, τόσο ώστε να μπορούν να μας ε, παρέχουν και ασφαλή τρόφιμα. Θα ε, δημιουργήσουμε λοιπόν προβλήματα για την ε, πάροχη υγιών τροφίμων προς τους καταναλωτές μας επειδή δεν υπάρχουν υποκατάστατες ουσίες για ορισμένες από αυτές που προτείνονται εδώ να απαγορευτούν. Και μάλιστα υπάρχουν στο πλαίσιο των κανόνων cut-off και πολύ συγκεκριμένοι αυστηροί περιορισμοί οι οποίοι εφαρμόζονται σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Κατά δική μου λοιπόν άποψη η τελική απόφαση που θα λάβει η Επιτροπή θα πρέπει να είναι εκείνη που θα καθορίσει κατά πόσο και ποιε από αυτέ τι ουσίε θα πρέπει να συνεχίσουν να ε, εγκρίνονται ή όχι. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό το αίτημα τη εισηγήτριας, δεν μπορούμε να προβέμουμε σε αυθαίρετες ε, ε, απαγορεύσεις συγγνώμη ουσιών, θα πρέπει να βασιστούμε σε επιστημονική αξιολόγηση όπω αυτή θα γίνει από την Επιτροπή. Ευχαριστώ σχολιάσατε μόνο το σημείο 6 και το σημείο 7 σήμερα σε και το Εφτακαλώς. Κύριε Βίζικ, σας παρακαλώ περιοριστείτε σε ένα λεπτό. Αλλά οι σοσιαλιστές, ε, το ID και οι πράσινοι δεν έχουν κάποιον πρόσωπο που θα πάρει το λόγο από τη δική τους πλευρά. Αυτό το ανακοινώνω προς ενημερωτικά για τους πολίτε. Κύριος Βίζικ, λοιπόν. Να σας ε, πω, Πρόεδρε, ότι ήμουν ως ε, σκιώδης ε, εισηγητής σε ένα σχετικό θέμα και αντιλαμβάνομαι πως το ζήτημα είναι περίπλοκο και δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε όλοι εύκολα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τις επιπτώσεις για την υγεία της χρήσης αυτών των ουσιών. Εγώ, λοιπόν, αυτή τη στιγμή θεωρώ ε, πως ε, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ε, για τους σοσιαλιστές τώρα. Δεν βλέπω να υπάρχει κανείς. Για το Ρινιού, δύο ομιλητέ. Μάρτιν Όψη και Ελέονορ Τριενό. Ποιος θα ξεκινήσει από τους δύο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αρχίζω εγώ και θα παρέμβω και για τις δύο αντιρρήσεις και θα με συμπληρώσει ο συνάδελφος. Μελέτησα λοιπόν προσεκτικά όλες αυτές τις ε, ουσίες. Έξι είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες και ξέρουμε τους κινδύνους, αναφέρθηκαν και πριν από λίγο μάλιστα. Ε, μία από αυτές τις ουσίες ε, δημιουργεί προβλήματα στο έμβριο, κάποια άλλη είναι ύποπτη για προβλήματα αναπαραγωγής και μια τρίτη ουσία έχει επισημανθεί από μία ομάδα καρκινολόγων. Τέλος, οι χρήστες που είναι γεωργοί υποβάλλονται οι ίδιοι σε μεγάλους κινδύνους για δερματοπάθειες. Μια άλλη ουσία επίσης είναι υπεύθυνη για νευρολογικά προβλήματα. Συνεπώς, η πιο βασική πρόληψη θα πρέπει να μας οδηγήσει να παρατείνουμε την απαγόρευση των ουσιών αυτών. 17 από αυτές έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο ε, σε πολλές ε, χώρες ε, που βρίσκονται σε στάση αναμονής για αυτές. Λοιπόν, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει κατάλογο ουσιών ανά είδος κινδύνου και όχι έτσι ένα μπέρδεμα ουσιών που όλες τις εξετάζουμε τον ίδιο τρόπο. Επίσης πρέπει να πιέσουμε τις χώρες μέλη που είναι υπεύθυνε για τις αξιολογήσεις ώστε να τις κάνουν τις αξιολογήσεις έγκαιρα μέσα στις προθεσμίες. Μία από τις ουσίες για παράδειγμα βρίσκεται σε μελέτη από το 2002, δεν έχει γίνει επαναξιολόγηση. Χτες άκουσα μία ευρωβουλευτή να λέει ότι τιμωρούμε τελικά τις ουσίες απαγορεύοντας τις. Εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρθα για να συνεισφέρω να σώσω ζωές και όχι να σώσω χημικά προϊόντα. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν είμαι κατά της παράτασης της ε, περίοδου έγκρισης των ουσιών αυτών και σήμερα το απόγευμα θα ε, ψηφίσω υπέρ της αντίρρησης που προτείνει η κυρία Χάζελκαμπ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Μάρτιν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η βάση της αντίρρησης είναι βέβαια η υγεία και το περιβάλλον και η προστασία τους από τα χημικά και δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε η συνάδελφος. Είναι σοβαρά αυτά που είπε και είναι πραγματικά ντροπή που έτσι μας φτάνει μια δέσμη χημικών ε, από τα οποία κάποια ε, προκαλούν ιδιαίτερες ανησυχίες, κάποια πολύ λιγότερες. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία, οι Ευρωπαίοι αγρότες, οι πολίτες, οι κατανοητές και το περιβάλλον. Εδώ μιλάμε για την πράσινη ανανέωση. Έτσι, εδώ βλέπουμε παλιά φυτοφάρμακα που γνωρίζουμε ότι πολλά από αυτά έχουν καταστροφικές συνέπειες, για παράδειγμα και στις μέλισσες όπως λέγαμε πριν, όχι μόνο στους ανθρώπους. Οπότε πώς είναι δυνατόν να τα αφήνουμε να κυκλοφορούν στην αγορά ενώ δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες, ενώ μπορούμε να βρούμε άλλες αναλλακτικέ φυτοφαρμάκων πολύ πιο ασφαλείς. Το σύστημα δεν ε, λειτουργεί. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις αντιρρήσεις και να δείξουμε ότι όχι απλώς πρέπει να παλαιγούμε από αυτά τα χημικά, ε, και φυτοφάρμακα, αλλά συγχρόνω πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξουν νέες μορφές περισσότερο ασφαλείς. Η κυρία Ριβαζή τώρα, εκ μέρου των Πρασίνων, τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ την κυρία Χάζενκαμπ για τις δύο αυτές αντιρρήσεις. Και εγώ θα αναφερθώ στο χλώρο τολερών και την φλουμιοξαζίνη. Ποια είναι τα κοινά αυτών των δύο ουσιών είναι ότι και δύο αυτές ουσίες έχουν ε, κατηγορηθεί ως ε, προτοξικές. Είτε πρόκειται για το χλωροτολινόν, είτε πρόκειται για την άλλη ουσία. Και στη συνέχεια ταξινομήθηκαν ως ε, δοκρινικοί διαταράκτες. Και έχουμε νόμους για τα φυτοφάρμακα, είτε πρόκειται ε, για τη μία κατηγορείται για την άλλη, είτε είναι προτοξικές, είτε είναι δηλαδή καρκινογόνες, είτε είναι ενδοκρινικοί διαταράκτε, πρέπει να απαγορεύονται. Τα ακούσαμε, υπάρχουν τοξικές επιπτώσει στην υγεία. Και τι κάνουμε εδώ και χρόνια, αναβάλουμε την αξιολόγησή τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Υπάρχει μια επιδημία καρκίνου στην Ευρώπη και ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στα φυτοφάρμακα, δεν λέω μόνο για τις δύο αυτές ουσίες, αλλά είναι ένα θέμα. Έχουμε και την κοινή γνώμη η οποία θέλει να σταματήσουν τα φυτοφάρμακα και εμείς τι κάνουμε. Καθυστερούμε, κολλησιεργούμε, λέμε να περιμένουμε άλλον ένα χρόνο για να γίνει εξολόγηση. Ε, λοιπόν, εγώ όταν κοιτάω το χλώρο διαπιστώνουμε ότι στο νερό υπάρχει υπέρβαση των ε, ποσοτήτων που επιτρέπονται και που οφείλεται αυτό στα φυτοφάρμακα. Και για την άλλη ουσία, την φλουμιοξαζίνη, εδώ ε, και χρόνια μιλάμε για την αντικατάστασή της λόγω τοξικότητας. Να τις εγκρίνουμε αυτές τις αντιρρήσεις. Ας πάψει πια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πάντα με τη βιομηχανία έχετε τους επιστήμονες, έχετε τις μελέτες που λένε ότι είναι τοξικές αυτές οι ουσίες και εσείς τι κάνετε, περιμένετε ακόμα επιπλέον μελέτες για να απαγορευτούν. Οπότε, ειλικρινά, πραγματικά εγώ στηρίζω αυτές τις δύο αντιρρήσεις και πρέπει να σταματήσουν αυτές οι ουσίες να κυκλοφορούν γιατί σκοτώνουν ανθρώπους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Δεν είσαι πικέ. Ταυτότητα και δημοκρατία δεν είναι εδώ. Για το ECR. Α, όχι, για το, ID, για το ECR. Για το ECR εγώ θα πάρω το λόγο. Παρακαλώ. Ωραία. Το ECR είναι κατά αυτών των αντιρρήσεων. Δεν πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπερβεί τι εκτελεστικέ τη αρμοδιότητε και τα μέτρα που προβλέπονται είναι απόλυτα συνεπή με τι νομικέ διαδικασίε, όπω αναφέρονται στην κυρία Πράξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δικιά τη τεχνική περίληψη είπε ότι οι παρατάσει που προβλέπονται είναι αναγκαίες γιατί δεν θα είναι δυνατόν να εγκριθεί ε, απόφαση για την ανανέωση όχι πριν εκπνεύσει η τωρινή άδεια. Και αυτά είναι εκτός ελέγχου από τους ετούντες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ε, καμία εξοδότηση των αρμοδιότητες για τις εκτελεστικές αυτές πράξεις. Και αν είμαστε κατά της παράτασης των 63 αυτών ουσιών, Έχουμε πόσες είναι, 44 στο πρώτο και 29 στο δεύτερο. Ε, τελικά απαγορεύουμε ουσίες οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και βρίσκονται στο τελικό στάδιο επαναξιολόγησης και επανέγκριση. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε έτσι. Ο κανονισμός έχει το καλύτερο σύστημα έγκρισης για τις δραστικές ουσίες και τα φυτοφάρμακα από παντού στον κόσμο. Γίνεται και αξιολόγηση, δημόσια διαβούλευση, συμπεράσματα από την ΕΦΣΑ, αποφάσεις από τη μόνιμη επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την ίδια την Εκτελεστική Επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να οδηγούν σε καθυστερήσεις όπως γίνεται τώρα. Οπότε, στις περισσότερες περιπτώσεις οι καθυστερήσεις αυτές δεν είναι ε, στα χέρια του ετούντα. Γι' αυτό και χρειάζεται αυτή η διαδικασία, ώστε να υπάρχει βεβαιότητα στην αγορά και προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι αγρότες και οι παραγωγοί έχουν τις ουσίες αυτές ως μέσα αντιμετώπισης ε, των ε, διαφόρων ασθενειών των φυτών. Λοιπόν, οι ουσίες αυτές όπως λέει το άρθρο 17 του κανονισμού 1107 και όπως είπε και η Ombudsman στην απόφαση 687 του 2018 η παράταση αυτή γίνεται κατανότατο για ένα χρόνο και απόφαση για την ανανέωση ή όχι της έγκρισης πρέπει να εγκρίνεται όσο γίνεται πιο γρήγορα. Συνεπώς, την περίπτωση που δεν υπάρξει ανανέωση της έγκρισης, ε, θα ανακληθεί η άδεια. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι οι παρατάσεις αυτές που αναφέρονται στην εκτελεστική πράξη δεν έχουν να κάνουν με ανησυχίες για την ασφάλεια των ουσιών αυτών. Αν υπήρχε κάποιος αρνητικός αντίκτυπος για την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων ή ε, καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, τότε θα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία κατά την οποία η μόνιμη επιτροπή θα είχε αποφασίσει διαφορετικά. Οπότε νομίζω ότι είναι ανόητο από την πλευρά μας να αντιτιθέμεθα στην έγκριση. Ευχαριστούμε. Πέντε λεπτά το πολύ θα πάρει το λόγο η Κομισιόν, η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ και θα μας ε, απαντήσει. Ε, η πρώτη μου ε, εμφάνιση είναι εδώ πέρα και έχει να κάνει μονίμως με αντιρρήσεις. Συμφωνούμε πλήρως ότι τα οικονομικά συμφέροντα δεν προέχουν όταν λαμβάνουμε αποφάσεις για φυτοφάρμακα. Λαμβάνουμε άπειρες επιστολές για το θέμα αυτό και παρόλα αυτά υιοθετήσαμε πολλές ε, ανακλήσεις. Ε, ή αρνηθήκαμε την ε, έγκριση πέρυσι. Δεν φοβόμαστε τη χημική βιομηχανία, δεν φοβόμαστε να πάμε τα δικαστήρια. Έχουμε 15 ε, υποθέσεις που τρέχουν ενώπιον τα, των δικαστηρίων και αυξάνει ολοένα ο ρυθμός. Επομένως δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτές οι παρατάσεις είναι απαραίτητες. Είμαστε υποχρεωμένε να τι δώσουμε με βάση το άρθρο 17 του κανονισμού PVP, φυτοπροστασίας δηλαδή, όπου λέει όταν η διαδικασία ανανέωσης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πέραν του, για λόγους πέραν του ελέγχου του ετούντα, η Κομισιόν πρέπει να παρατείνει την περίοδο έγκρισης. Δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουμε κάτι άλλο και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον διαμεσολαβητή, όπως ανέφερε και η κυρία Μάκεντάιρ. Ο λόγος για τον οποίο καθυστερήσαμε είναι συνήθω ο κλασικό, γιατί τα κράτη-μέλη δεν δίνουν ε, εγκαίρω εκθέσει του. Και αυτό το τόνισε ε, και κάποιοι ευρωβουλευτέ. Ε, ένα ο φάκελος υποβλήθηκε από στις 30 Απριλίου του 2015 στη Γαλλία και θα έπρεπε να είχαν δώσει την έκθεσή του σε ένα χρόνο μετά, τον Απρίλιο του 2016. Ε, δόθηκε στην ΕΦΣΑ μόλις τώρα. Τρία χρόνια καθυστέρηση από τον εισηγητή και τον συνεισηγητή για να ετοιμάσουν την έκθεση. Αυτό, γι' αυτό δεν φταίει ο ετών. Επίσης, να, να αντιδράσω σε ένα από τα στοιχεία που είπατε. Το δικαστήριο, ή μάλλον υπάρχουν τα, συμφωνούμε με τα ενδιάμεσα κριτήρια, Επίσης, το Μάρτιο φέτο ε, συμφωνήθηκε ότι το ράκ δεν θα πρέπει να θεωρηθεί τοξικό. Έχει αλλάξει πρόσφατα λοιπόν η κατάσταση. Το άρθρο 17 δεν μας αφήνει περιθώριο ελιγμών δυστυχώς. Εάν διαδικασίες δεν ολοκληρωθούν για λόγους πέραν του ελέγχου του ετούντα και δεν έχουμε σαφή ένδειξη ότι τα κριτήρια ε, έγκρισης δεν πληρούνται, θα πρέπει να δώσουμε παράταση. Βεβαίως, Υπάρχει το εξή με το Κοινοβούλιο. Αν κατά την αξιολόγηση των, ε, του peer review υπάρχουν ε, ε, ενδείξεις ότι τα κριτήρια δεν πληρούνται και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, προτείνουμε για πρώτη φορά να ανακαλέσουμε την ε, έγκριση γιατί υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από τις ουσίες που υπάρχουν εδώ στους δύο κανονισμούς. Εδώ δεν είμαστε στη φάση όπου έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι τα κριτήρια έγκρισης δεν πληρούνται. Έτσι, αυτό είναι διαφορετικό. Είναι μια άλλη υπόθεση που θα τη συζητήσουμε σήμερα στην Επιτροπή Άκρη το απόγευμα. Ε, Δυστυχώ είμαι σε αυτή τη φάση. Λυπόμαστε που τα κράτη-μέλη δεν έχουν κάνει τη δουλειά του εγκαίρω και θα το αντιμετωπίσουμε και στην ε, αξιολόγηση ρήφη του κανονισμού, είναι ένα από τα μείζωνα προβλήματα ότι τα κράτη-μέλη δεν σέβονται τις προθεσμίες και δεν ολοκληρώνουν το έργο τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Ευχαριστώ, πολύ. Θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα για τις αντιρρήσεις αυτές. Θα έχουμε ως τα αποτελέσματα. Και περνάμε τώρα στην άλλη συζήτηση πριν από τις ε, ψηφοφορίες του απογεύματος για τρεις αντιρρήσεις για μη, μη γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, κοινή συζήτηση πάλι. Τρεις αντιρρήσεις λοιπόν. Θα τις συζητήσουμε μαζί. Τιλιμέτ, εισηγητής. Πασκάλ Κοφά. Yes, uh, we are Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ναι, εδώ αναφερόμαστε σε αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά ε, γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο σόγια και αραβόσιτο ε, και συγκεκριμένα τέσσερα συμβάντα αραβοσίτου και τις 14 του 14 συνδυασμού αυτών των συμβάντων στον Αραβόστο. Γιατί έχουμε λοιπόν ε, προβεί σε αυτή την εισήγηση. Καταρχήν, δεν υπήρξε δημοκρατική διαδικασία στην ε, λήψη των αποφάσεων και δεν γνωρίζουμε τι λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόψη τη όταν λαμβάνει τι ειδικέ αποφάσει. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά του κινδύνου ε, για την υγεία των ανθρώπων, μιλάμε εδώ για ε, ε, κάποια, κάποιες καλλιέργειες οι οποίες έχουν τροποποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχουν αντοχή, ανθεκτικότητα σε περισσότερα από ένα προϊόντα φυτοπροστασίας. Ε, και παρότι το κάνουμε ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά αυτό οδηγεί ε, στην υπερβολική χρήση των, των φυτοφαρμάκων όπως για παράδειγμα της γλυφοζάτης. Δηλαδή, ε, ποια είναι η αντίδραση από την πλευρά των ε, ε, των, εταιρείων που κατασκευάζουν φυτοφάρμακα να χρησιμοποιούν ακόμα περισσότερα φυτοφάρμακα αφού υπάρχει υψηλότερη ανθεκτικότητα αυτών των επικοιλίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσει στο περιβάλλον, στη βιοπικιλότητα, στην υγεία των καταναλωτών και εδώ αναφέρομαι γενικότερα και στι εισαγωγέ τροφίμων και ζωοτροφών. Ε, γνωρίζουμε ότι η γλυφοσυνάτη και η γλυφοζάτη είναι τα, ε, οι ουσίε τι οποίε ακριβώ έχουν δημιουργηθεί ποικιλίε για να είναι ανθεκτικέ. Αλλά η γλυφοσυνάτη δεν χρησιμοποιείται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και τοξική για την αναπαραγωγή. Ε, και γνωρίζουμε ε, τα, όλα τα επιστημονικά δεδομένα σε ό,τι αφορά την δημιουργία καρκίνου λόγω τη γλυφοσάτη. Οπότε δεν αντιλαμβανόμαστε το γιατί δεν λαμβάνει υπόψη η ΕΦΣΑ τις επιπτώσεις από τον ψεκασμό με συμπληρωματικά φυτοφάρμακα αφού ουσιαστικά εδώ έχουμε ένα κοκτέιλ διαφορετικών φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται ε, σε σχέση ακριβώς με τέτοιου είδους γενετικά τροποποιημένα ε, φυτά. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν τέτοιου είδους δοκιμές ασφαλείας, χρειάζεται να επιστρέφουμε στις λεπτομέρειες και όχι απλώς να εξετάζουμε ε, τον ε, γενετικά τροποποιημένο οργανισμό, το φυτό αυτό κάθε αυτό. Και μετά σε ό,τι αφορά τον αραβόσιτο που έχει περισσότερες από μία τροποποιήσεις, περισσότερα από συμβάντα, περιλαμβάνει και αντοχή στο BT toxin όπως λέγεται, αλλά εδώ δεν έχει γίνει μία δοκιμή, μία εξέταση από την ΕΦΣΑ κατά ως προς το ποιε είναι οι επιπτώσεις αυτών των τοξινών BT. Οπότε δεν μπορούμε, αυτό είναι το σκεπτικό μας, να επιτρέψουμε αυτούς τους, ε, αυτά τα γενετικά τροποποιημένα φυτά χωρίς να γνωρίζουμε τις ακριβείς τους επιπτώσεις για το περιβάλλον, για τα ίδια τα φυτά και για τους ανθρώπους. Δεύτερο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Ε, το θυμάμαι, ε, γιατί με ε, ένα συναδελφός, ότι αναφέρθηκε ότι υπήρξαν 36 διαφορετικές αντιρρήσεις ε, που εκφράστηκαν από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και δεν υπήρξε καμία ειδική πλειοψηφία που να συγκεντρώθηκε σε επίπεδο κρατών μελών. Παρόλα αυτά όμως τελικά δόθηκε έγκριση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ουσιαστικά λοιπόν δεν υπάρχει δημοκρατική διαδικασία σε ό,τι αφορά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Ερωτώ λοιπόν την Επιτροπή, γιατί συνεχίζει λοιπόν να εγκρίνει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς όταν δεν έχει ε, λάβει την υποστήριξη ούτε από Ούτε τα κράτη-μέλη, από το Συμβούλιο, ούτε από το Κοινοβούλιο το οποίο εκφράζει τη βούληση των πολιτών. Και ένα τρίτο επιχείρημα ε, που θα ήθελα να θέσω εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα του τι λαμβάνεται ακριβώς υπόψη στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, ποιοι είναι δηλαδή οι, οι θεμητοί εκείνοι λόγοι κατά την άποψη της Επιτροπής που την οδηγούν στο να λάβει αυτή την απόφαση όταν δεν υπάρχει υποστήριξη ούτε από το Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο και τι κάνει ε, σε σχέση ακριβώς με τα όσα έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων, ε, των, ε, της ε, Σύμβασης των ΗΠΑ για τη Βιοπικιλότητα, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Όλε αυτέ λοιπόν οι διεθνείς συμφωνίε τι οποίε έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν κανένα βάρο, δεν έχουν καμία σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έχει να μα πει και να σα πω κάτι σε σχέση σε ό,τι αφορά με τη σόγια εδώ, τη γενετικά τροποποιημένη σόγια. Ουσιαστικά πρόκειται για μία από τι κύριε καλλιέργειε που χρησιμοποιείται και οδηγεί σε αποψήλωση των δασών. Δεν θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούνται τέτοιου είδου καλλιέργειε αν οδηγούν στην αποψήλωση. Και από εκεί και μετά ε, πέρυσι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μία έκθεση σε ό,τι αφορά την αποψήλωση των δασών και σε δική της ανακοίνωση πρόσφατη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στην ανάγκη του να λάβουμε περισσότερες δράσεις ούτως ώστε να προστατεύσουμε τα παγκόσμια δάση. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν πώ ε, συνάδει κάτι τέτοιο με τι απόψει τη Επιτροπή. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ακούσω τι απόψει αλλά και να λάβω την υποστήριξή σα ε, για αυτό το αίτημά μα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Θα δώσω τώρα το λόγο στι πολιτικέ ομάδε. Η κυρία Μπογιάν τώρα για το ΕΛΚ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ενημερώθηκα ότι είχαν τεθεί πολλέ αντιρρήσει κατά την προηγούμενη βουλευτική θητεία και βλέπω να υπάρχουν πολλέ τέτοιε αντιρρήσει να συνεχίζονται. Ε, Χωρί να υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα, η ΕΦΣΑ έδωσε το πράσινο φω για αυτού του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, χωρί όμω να γνωρίζουμε αν είναι πιο επιβλαβεί από τι συμβατικέ αντίστοιχε επικοινίε. Εάν η ΕΦΣΑ εμ, όμως θεωρεί ότι πράγματι ένα προϊόν είναι εμ, ασφαλές, ε, τότε θα πρέπει να εμπιστευόμαστε την δική της εμπειρογνωμοσύνη. Αυτή είναι η κανόνες επί των οποίων έχουμε συμφωνήσει και δεν θεωρούμε κατά συνέπεια ότι έχουν εμ, υπερβεί ε, τις αρμοδιότητες, τις, τις αρμοδιότητες, αρμοδιότητες συγγνώμη, τους οι συνάδελφοί της ΕΦΣΟ. οπότε θα ήθελα ε, να καλέσω τους συναδέλφους να καταψηφίσουν αυτή την πρόταση. Για τους σοσιαλιστές τώρα, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Σίλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Ε, τα τρία προηγούμενα ψηφίσματα και προτάσει ε, που γίνονται ε, σε ό,τι αφορά την απαγόρευση αυτών των γενετικά τροποποιημένων ε, ποικιλιών αραβοσίτου, σόγια και άλλων, έχουν λάβει την υποστήριξη από τρει διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε και νομίζω πω με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε και ένα ισχυρό μήνυμα κατά την έγκριση. Γιατί ο στόχο μα θα πρέπει να είναι καμία έγκριση γενετικά τροποποιημένων φυτών και άλλων οργανισμών εφόσον δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται σε ό,τι αφορά τι δυνητικέ επιπτώσει στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Και βέβαια το ερώτημα που τίθεται είναι το τι θα κάνει στο μέλλον η Επιτροπή με τι αποφάσει που λαμβάνουμε πλειοψηφικά εδώ στο Κοινοβούλιο. Η νέα πρόεδρο τη Επιτροπή είπε ότι από εδώ και στο εξή θα σέβεται περισσότερο αυτέ τι πλειοψηφικέ αποφάσει του Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδου καταστάσει στο μέλλον εδώ στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ. Thank you. So for... Ευχαριστούμε η κυρία Δανούτα. Ο κύριο Ταντάβαρ. Το Ρινιού. Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να είναι ιδεολογική αυτή η συζήτηση για το κατά πόσο στηρίζουμε ή όχι τα γενετικά τροποποιημένα. Πρέπει να βασιζόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα. Εγώ έχω συνυπογράψει δύο από τι τρει αντιρρήσει για ε, συγκεκριμένου λόγους. Πιστεύω ότι τα γενετικά αυτά τροποποιημένα είναι για να είναι πιο ανθεκτικά στα φυτοφάρμακα. Ε, το ένα έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο ακόμα συζητάμε τις γενικές ιδιότητες. Θα κινδυνεύαμε να αυξήσουμε τα χημικά και τα φυτοφάρμακα ε, από την πίσω πόρτα με τη διαδικασία αυτή. Επιπλέον, αυξάνεται και η αντίσταση των ζυζανίων στα φυτοφάρμακα. και έτσι υπάρχει κίνδυνος για την επόμενη γενιά. Συνολικά η ομάδα μας, ξέρετε, είναι υπέρ της καινοτομίας, είναι υπέρ του να έχουμε μια σωστή και σοφή προσέγγιση, αλλά εδώ δεν πρόκειται για την ε, καινοτομία, γιατί για 10 χρόνια δεν έχει υπάρξει τίποτα καινούργιο με καινοτομία από την κυκλοφορία αυτών των προϊόντων όπως ε, βλέπουμε και στο άρθρο 168 της συνθήκης. Διάφορες πολιτικές ομάδες έχουν συνυπογράψει τις αντιρρήσεις αυτές και έχω και ένα θεσμικό ερώτημα. Είπατε ότι στην προηγούμενη περίοδο υπήρχαν δεκάδες και δεκάδες τέτοιες αντιρρήσεις. Λοιπόν, αναρωτιέμαι, μήπως θα μπορούσαμε να δουλέψουμε παραπάνω στην νομική βάση και να μην έχουμε να κάνουμε μόνο με εκτελεστικές αρμοδιότητες αλλά και σε κατεξουσιοδότηση πράξης. Είναι νομίζω ο καλύτερος τρόπος, ο μόνος τρόπος για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Θα ήθελα τη γνώμη σα ή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μήπως αντί για τις εκτελεστικές πράξεις περάσουμε στις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε, ε, συγγνώμη, η Επιτροπή μας ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει την νομοθεσία και να προτείνει μια νέα. Οπότε τώρα το μπαλάκι είναι ε, στα χέρια της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τη Δευτότητα και δημοκρατία δεν έχουμε κανέναν. Α, εσείς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορεί να έχουμε 60.000 ε, σόγια από τη Βραζιλία στη Γαλλία πριν από λίγο, αλλά σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των εισαγωγών σόγια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος ε, εισαγωγέας ε, σόγιας από την Βραζιλία, κυρίω που είναι και γενετικά τροποποιημένη. Και το παράδοξο είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρε απαγορεύουν να παράγεται στο έδαφο του γενετικά τροποποιημένη σόγια, ενώ την εισάγει απ' έξω, μαζικά μάλιστα. Σύμφωνα με την ε, Greenpeace της Γαλλίας, η Ευρώπη και κυρίως η Γαλλία δεν χρειάζεται να εισάγει τέτοια προϊόντα από την άλλη άκρη του κόσμου. Ο κύριος Μακρόν εξάλλου είχε πει ότι ήθελε μια πρωτεϊνική κυριαρχία της Ευρώπης. Να έχει δηλαδή αρκετές ε, πρωτεΐνες από μόνη της Ευρώπη και ίσως θα μπορούσε να αντικατασταθεί σόγια από άλλη φυτική πρωτεΐνη, ολική ε, και κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δεν θα έπρεπε να επιμένει στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που τελικά οδηγούν σε καταστροφή το περιβάλλον. Ευχαριστούμε. Για το ECR, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε κατά όλων των αντιρρήσεων αυτών εμείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υπερβεί τις εκτελεστικές της εξουσίες και τα σχέδια που προτείνονται συνάδουν πλήρως με την νομική διαδικασία που αναφέρεται στη βασική πράξη. Η διαδικασία αξιολόγησης των καλλιεργών αυτών που έχουμε στην Ευρώπη είναι από τις πιο αυστηρές. Επιτρέπει στις χώρες μέλη και στο κοινό να παρεμβαίνουν να ενημερώνονται και είναι αρκετά ισχυροί ώστε να μπορούμε να πούμε ότι τα γενετικά προϊόντα που εγκρίνονται είναι εξίσου ασφαλή όσο και τα άλλα, τα συμβατά. Και πρέπει να ακούμε την επιστήμη. Έχουν γίνει ανεξάρτητες ε, μελέτες και θα έπρεπε να υπάρχει πρόσβαση σε αυτές. Αν εξακολουθούμε να ε, αμφιβάλλουμε για την ε, γυρότητα και την ε, ουδετερότητα της επιστήμης τότε που πάμε. Στην τελευταία θητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προφορικές ερωτήσεις και ψήφισμα για την, ε, τον δισταγμό που έχει το κοινό στον εμβολιασμό. Πώ είναι δυνατό όμω να επικρίνουμε αυτού που δεν εμβολιάζουν τα παιδιά του όταν χρησιμοποιούν επιστημονική γνώση, ενώ συγχρόνω αγνοούμε τα συμπεράσματα οργάνων όπω είναι η ΕΦΣΑ, που λέει ότι οι γενετικά τροποποιημένε καλλιέργεια είναι απόλυτα ασφαλής. Επίσης, αφισβητούμε ε, τα επιχειρήματα στις αντιρρήσεις αυτές ε, για την χρήση τη γλυφοσάτης και της γλυφοσινάτης, διότι δεν λαμβάνουν υπόψη την αδειοδότηση. Και δεν είναι σωστό να γίνεται η σύνδεση αυτή. Εμείς έχουμε επίπεδα ανώτατα για τα υπόλοιπα από τις ουσίες αυτές και δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι διαφορετικό για τα μη γενετικά ε, προϊόντα. και νομίζω ότι το πάνελ της ΕΦΣΑ σε όλες τις περιπτώσεις δεν εντόπισε καμία ανησυχία όσον αφορά την κατανάλωση από τον άνθρωπο για την τοξικότητα και την δυνατότητα ε, παρουσίασης ε, αλλεργιών. Εξαρτάται η Ευρώπη από τις καλλιέργειες σόγιας, πρωτεΐνης σόγιας, για τις ζωοτροφές. Οπότε η διαδικασία έγκρισης πρέπει να ολοκληρώνεται όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε να μην μένουμε σε καθυστέρηση σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και να διατηρήσουμε τον ανταγωνισμό μας στο διεθνές εμπόριο. Ε, από την ΚΟΕ. Καίγεται ο Αμαζόνιος. Πολύ περισσότερο παραποτέ. Και η οργή κατά της αποψήλωσης ε, εναντίον ε, αυτού, ε, για αυτό το πολύτιμο οικοσύστημα είναι όλο και μεγαλύτερη. και όμως η Κομισιόν επιτρέπει γενικά τροποποιημένη σόγια και καλαμπόκι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι προφανή όλα, όλες τα, για όλους. Ε, αποψηλώνται τα δάση στον Αμαζόνιο για να παράγουμε, ε, για να καλλιεργήσουμε σόγια αραβόσιτο και να παράγουμε ε, φτηνά ε, προϊόντα. Ε, χρησιμοποιούνται αυτές οι ποικιλίε για τις οποίες έχουμε αντίρρηση. Η Κομισιόν ξέρει ότι αυτές οι γάμματα φόμικρον ε, είναι ανθεκτικές στη γλυφοσάτη και γλυφοσυνάτη. και χρησιμοποιείται μια ε, γεωργία που προκύπτει από την ε, κρίζωση και την ε, καύση της γης, ας πούμε. Πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση κρέατος, το ξέρετε, το ξέρετε για να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος. Ξέρετε ότι κινδυνεύει ο πληθυσμό στι χώρε εξαγωγών και αυτά τα προϊόντα μπαίνουν στι αγορέ μα επίση. Η Κομισιόν ξέρει ότι δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση στις εγκρίσεις αυτών των γαμματάφα όμικρων. Ε, τουλάχιστον θα έπρεπε να το ξέρει. Γιατί λοιπόν δεν σταματάτε αυτή την α, ανεύθυνη συμπεριφορά, αυτή τις ανεύθυνες εγκρίσεις. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν για πέντε λεφτά το πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι. Χαίρομαι που συναντάω το νέο κοινοβούλιο, τη νέα, τη νέα επιτροπή σας, παρότι βλέπω αντιρρήσεις εναντίον θέσεων της Κομισιόν. Θέλω να σα εξηγήσω πώ εφαρμόζουμε την νομοθεσία και προστατεύουμε την ανθρώπινη ε, υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον. Μιλάμε για δύο εγκρίσει ε, γαματαφόμικρων και μία ανανέωση τη όγια ε, που είναι ήδη στην αγορά. Συνοψίζω πολύ σύντομα. Η ΕΦΣΑ έκανε μία πολύ πλήρη αξιολόγηση κινδύνου και συμμορφώθηκε με τους κανόνες στον κανονισμό και με την αξιολόγηση κινδύνου, τις κατευθυντήρες για την αξιολόγηση κινδύνου της ΕΦΣΑ. Και δεν υπήρξαν καθόλου δεδομένα ε, που έδειξαν το αντίθετο. Επίσης, τα κράτη-μέλη σχολιάζουν το έργο της ΕΦΣΑ. Η ΕΦΣΑ κοίταξε όλα τα σχόλια και απάντησε στα κράτη-μέλη και όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΦΣΑ. Υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις κριτικές που άσκησαν τα κράτη-μέλη ή αμφισβήτησαν κάποια επιστημονικά στοιχεία. Τα σχόλια και οι απαντήσεις της ΕΦΣΑ είναι τμήμα της νομοδότησης της ΕΦΣΑ. Επίσης σημαντικό, σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα, οι αδειοδοτήσεις, οι εγκρίσεις για τις οποίες μιλάμε αφορούν τις εισαγωγές. Η καλλιέργεια γίνεται σε τρίτες χώρες και τα φυτοφάρμακα και ζυζανιοκτώνα ψεκάζονται σε τρίτες χώρες. Σημαντικό. Επίσης, όταν τα προϊόντα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι γάματα φόμικρον, είτε είναι συμβατικά προϊόντα, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα μέγιστα όρια καταλήπων. Και τα μέγιστα όρια καταλήπων καθορίζονται στον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα που επίσης ε, καλύπτει και αυτά τα προϊόντα. Επομένω, η προστασία τη ανθρώπινη υγεία εξασφαλίζεται μέσω του σεβασμού των μέγιστων ορίων καταλήπων. Τώρα για την αντίληψη του κόσμου, για τις απόψεις του κόσμου, του κοινού. ο κόσμος έχει δυνατότητα να σχολιάσει την γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ και η ΕΦΣΑ απάντησε με διαφανή τρόπο σε όλα τα σχόλια που έκανε το κοινό. Η ΕΦΣΑ κατέληξε ξεκάθαρα ότι είναι ασφαλή αυτά τα προϊόντα για την ανθρώπινη υγεία, για την υγεία των ζώων και για το περιβάλλον. Με βάση τα στοιχεία αυτά, υποβάλαμε τις προτάσεις στις επιτροπές των κρατών μελών που θα πρέπει να ψηφίσουν για τις αποφάσεις αυτές. Και κυρίως για πολιτικούς λόγους τα κράτη-μέλη δεν πήραν θέση. Δεν ήταν κατά, ούτε υπέρ όμως. Αυτά στη μόνιμη επιτροπή, έτσι, και μετά στην Επιτροπή Προσφυγών. Με όλα αυτά τα δεδομένα υπάρχει νομική υποχρέωση για την Κομισιόν υπό την νομοθεσία για τους γάμα τάφο μικρών να λάβει απόφαση. Η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ είναι θετική για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον. Είναι καθήκον τότε της Κομισιόν να υιοθετήσει τις αποφάσεις έγκρισης. Σε ό,τι αφορά την επιτροπολογία και τη δημοκρατία που σχολιάσατε μερικοί ομιλητέ, φυσικά η Κομισιόν θα ήθελε να εισαγάγει περισσότερη δημοκρατία. Και υπάρχει μια πρόταση η οποία συζητείται αυτή τη στιγμή. Μέχρι όμως να υιοθετηθεί αυτή η, η πρόταση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ε, συμμορφωθούμε τους κανόνες και να εφαρμόσουμε τους κανόνες. Με όλα αυτά, και ε, τα λέω όλα αυτά, διότι τα, το δεδομένο είναι ότι η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ είναι θετική. Ε, η νομοθεσία για την φυτοπροστασία λέει ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τα μέγιστα όρια καταλήπων. Σε ό,τι αφορά την ε, ανεξαρτησία ή μάλλον την εξάρτηση από Τροφέ και ζωοτροφέ που εισάγονται από τρίτε χώρε. Είναι πολύ ψηλή και θέλουμε να μειώσουμε αυτή την εξάρτηση. Σωστό είναι, αλλά υπάρχει. Και χρειαζόμαστε αυτού του σπόρους σόγιας για τη γεωργία μα και για τη διατροφή μα. Ε, υπάρχει αγορά που ζητάει αυτά τα προϊόντα. Εάν η αγορά δεν τα ζητούσε, ακόμα και αν τα εγκρίναμε, δεν θα τα εισαγάγαμε, διότι κανένα δεν τα αγόραζε. Επομένω, καταλήγω ότι σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότηση ακολουθήσαμε όλα τα βήματα με διαφανή τρόπο σεβόμενη την νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά την εξάρτηση από τις εισαγωγές και σε ό,τι αφορά το θέμα της σύμβασης του ΟΗΕ και άλλων διεθνών συμφωνιών, φυσικά αυτά είναι θέματα σημαντικά. Και η Κομισιόν εφαρμόζει όλες αυτές τις συμβάσεις και συμφωνίες, αλλά δεν συνδέονται άμεσα με τις εγκρίσεις τις οποίες συζητάμε σήμερα. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ που μας δώσετε το λόγο και ελπίζουμε να συνεχίσουμε επικοδομητικό διάλογο και στο μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα κλείσουμε αυτή τη δεύτερη συζήτηση της πρωινής συνεδρίασης και θα τα ξαναπούμε στις 2.30 το απόγευμα και μετά θα ψηφίσουμε. Μην ξεχάσετε τις κάρτες ψηφοφορίας σας γιατί θα ξεκινήσουμε πάρα αυτά με ψηφοφορία και δεν θα έχετε χρόνο να πάτε στο γραφείο σας. Ε, θα, θα σας ξαναδώ το απόγευμα.